As Δεδομένου ότι μόνο μία ώρα έχουμε για να συζητήσουμε δύο εκθέσεις, θα ήθελα να ξεκινήσουμε. Λυπάμαι για αυτούς που έχουν αργήσει, δεν μπορούμε να τους περιμένουμε όλους. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την έκθεση για την εξέλιξη των μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο εισηγητής είναι ο Φρανσουά Αλφονσί και θα του δώσω το λόγο απευθείας να κάνει τις εισαγωγικές παρατηρήσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, με δύο λόγια θα σας παρουσιάσω το έγγραφο που ήδη έχουν πάρει όλα τα μέλη της Επιτροπής που αφορά στην ε, εξέλιξη και την μακροπεριφερειακή στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η οποία ασχολείται με κυρίως με τη Μεσόγειο. Η μακροπεριφερειακή στρατηγική στην Ευρώπη είναι πρόσφατη διαδικασία. Η πρώτη μακροπεριφέρεια δημιουργήθηκε το 2009 στη Βαλτική. Η ιδέα αυτού του νέου ε, πεδίου δημόσιας ευρωπαϊκής πολιτικής ε, αφορά μια περιοχή η οποία έχει τα χαρακτηριστικά συνεκτικής ε, περιφέρειας στα πλαίσια μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής στη Βαλτική με τέσσερις, ε, με τέσσερις ε, πυλώνες και τέσσερις άξονες προτεραιότητες. Μετά την ε, Βαλτική και η, περιφέρεια του, και η περιοχή του, του Δούναβη ξεκίνησε μια τέτοια μακροπεριφέρεια που ασχολείται με την ίδια υδατική λεκάνη μέσα στο ίδιο, ανάμεσα στους ίδιους ορεινούς όγκους την, ανάπτυ... την ε, πρόθεση μιας ε, περιφερειακής πολιτικής, δίκτυα και μια ολοκληρωμένη ε, θαλάσσια πολιτική. Έτσι για μας η μακροπεριφερειακή πολιτική ανοίγει νέες προπτικές στο επίπεδο της εδαφικής συνεργασίας που είναι η τρίτη ε, πολιτική, τρίτη προτεραιότητα ε, στην πολιτική συνοχής. Έτσι λοιπόν μετά από αυτή την πρώτη εμπειρία αποφασίσαμε να δούμε τα αποτελέσματα και τι διαπιστώνουμε. Υπάρχει καταρχήν μια συγκεκριμένη προσδοκία για να ασχοληθεί κανείς με αυτό το νέο πεδίο δημόσιας πολιτικής στην Ευρώπη με βάση την ε, ανάπτυξη σε εδαφική, σε μια συγκεκριμένη εδαφική περιοχή ε, προωθεί την ευρωπαϊκή εξέλιξη, επιτρέπει στους Ευρωπαίους που μοιράζονται την ίδια περιοχή, που έχουν κοινή ιστορία, να ενισχύσουν ή να αποκαταστήσουν καμιά φορά τους δεσμούς τους και να ξεκινήσουν σε κοινή βάση την ανάπτυξη. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε έκθεσή της τον Ιούνιο του 2011 υπογράμμισε το πόσο ενδιαφέρουσα είναι αυτή η μακροσυνεργασία και βεβαίω η χρηματοδότηση αυτών των περιοχών με βάση τους στόχους. Ασχολήθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε μια στρατηγική για την Βαλτική και στην ε, περίπτωση του Δούναβη και πάλι ε, κλήθη από το Συμβούλιο να παίξει τον ρόλο της κινητήριας δύναμης σε αυτή τη στρατηγική. Βεβαίω όμω πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η διακυβέρνηση ενό τόσο σύνθετου ε, εργαλείου απαιτεί σημαντική τεχνική βοήθεια και αυτή τη στιγμή η Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο μας είπε ότι δεν μπορεί να αναλάβει κάτι περισσότερο όσο έχουν τα πράγματα. Από την άλλη πλευρά ε, η εμπειρία που έρχεται από αλλού η εμπειρία επίσης δείχνει ότι δεν μπορεί μια μακροπεριφέρεια να μην έχει πραγματική αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό το Συμβούλιο ε, κατέληξε σε ένα, συμβούλιο, σε ένα κανόνα των τριών όχι όπως ονομάστηκε δηλαδή σε, μη, σε όχι σε νέες χρηματοδοτήσεις, όχι σε νέο ρυθμιστικό πλαίσιο κλπ. Αλλά στις 13 ε, του περασμένου Απριλίου, την διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας, το Συμβούλιο ναι, άλλαξε και ε, κατέληξε στον κανόνα των τριών ναι, ε, Δηλαδή ναι στη συμπληρωματικότητα των χρηματοδοτήσεων, ναι στο συντονισμό των θεσμικών οργάνων, ναι στον καθορισμό νέων σχεδίων. Η συγκεκριμένη διαλεκτική επιδιώκει ουσιαστικά την αναζήτηση μιας κατάλληλη ισορροπία που πρέπει να προσδιοριστεί πριν από την οριστική θέσπιση των κανονισμών της προσεχούς Πολιτική Εδαφική Συνοχή για την περίοδο 2014-2020. Οπότε μπορεί κανείς να υπογραμμίσει την υπεραξία της μακροφερειακής στρατηγικής. Μέσω από το, του παραδείγματος της Βαλτικής θάλασσας αναδεικνύονται αρκετές δυνατότητες χάρη στην εφαρμογή μακροφερειακών στρατηγικών. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για την παροχή ενός κατάλληλου πλαισίου αναφοράς στις πολιτικές συνοχής και τη διευκόλυνση της διατομεακής συνεργασίας σε μια δεδομένη κοινότητα. Αυτό το πλαίσιο δίνεται να προσανατολίσει επενδύσεις και χάρη στη συνολική εικόνα υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας πραγματικών συνεργειών. Ένα άλλο πλεονέκτημα της εν λόγος στρατηγική στρατηγικής και άλλη προστιθέμενη αξία είναι ότι επιτρέπει μεγαλύτερη συμμετοχή και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων μέσων παρέμβαση που έχει στη διάθεσή της η Ένωση, όπως ας πούμε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης επιτρέπει τη σύγκληση μεταξύ των πόρων των περιφερειών, των κρατών μελών και των Ευρωπαϊκών Ταμείων μέσω μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Ε, όλοι θεωρούν ότι η σύγκληση των πόρων με αυτόν τον τρόπο είναι μια στρατηγική που είναι υποφελής για όλους. Η μακροπεριφερειακή στρατηγική ε, στο πλαίσιο της ε, πολιτικής γειτονίας μπορεί να διευκολύνει και να είναι παραγωγική. Αυτό είναι η προστιθέμενη αξία που προκύπτει. Τώρα, οι δυσκολίες. Φυσικά όλα αυτά δεν γίνονται μόνα τους Πρώτη δυσκολία είναι ότι κάθε μακρο, μακροπεριφέρεια έχει διπλή διάσταση. Μία εδαφική, λόγω του προσδιορισμού ενός κατάλληλου δαφικού πλαισίου εφαρμογής και μια λειτουργική διάσταση μέσω του καθορισμού των προτεραιοτήτων. Η, αυτή η διπλή διάσταση δεν μπορεί να επιτευχθεί αυθόρμητα ευθύς εξ αρχής Όλα αυτά τα στάδια ε, απαιτούν ένα εκ των προτέρων σχεδιασμό. Και ε, η διάρκεια αυτή, ε, η διάρκεια της θα είναι ενός ή δύο ετών. Πρέπει λοιπόν να καθοριστούν οι προτεραιότητες που θα αποφασίσει να έχει αυτή η μακροπεριφέρεια. Η λειτουργία των μακροπεριφερειών πρέπει να προκύπτει από πρέπει να αποφύγει την παγίδα της διακυβερνητικής διακυβέρνησης, αλλά να, να μην περάσει προς το διακυβερνητικό και να ε, προτιμήσει μια ε, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που θα δίνει έμφαση στο περιφερειακό επίπεδο. Γιατί, Γιατί αυτό εξασφαλίζει ότι θα έχουμε μια ευρωπαϊκή αποστολή, μια ε, μια ε, ε, κατεύθυνση προς περιφερειακή ανάπτυξη σύμφωνα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ο σχηματισμός των μελλοντικών μακροφεριών δια της αυθόρμητης δημιουργίας δεν μπορεί να αποτελέσει τον τρόπο που θα προχωρήσουμε. Υπάρχει ένα στοιχείο τυχαίο το οποίο δεν θα είναι θετικό για την ανάπτυξη συνεκτικών δράσεων. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ξεκινήσει εκ των κάτω. Τέλος, η συμμετοχή των περιφερειών της γειτονίας είναι απαραίτητη για την έγκριση πολλών σχεδίων που εντάσσονται στο πλαίσιο των μακροπεριφερειακών στρατηγικών, όμως πρέπει να προκύπτει από τις εδαφικές πολιτικές και να μην αποτελεί ε, συνιστόσα κάποιας εξωτερικής πολιτικής, η οποία δεν είναι κατάλληλη για τις ε, ε Τι πρέπει να γίνει για να ληφθούν υπόψη αυτά τα πρώτα συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι η μακροπεριφερειακή πολιτική πρέπει να ενταχθεί στα πλαίσια μιας συνολικής πολιτικής για να μην έχουμε απλώς θέματα άμεσης πολιτικής να μας απασχολούν. Δηλαδή, ένας χάρτης προβλέψεων των ευρωπαϊκών μακροφεριών που θα μπορούσε να συνταχθεί και θα είναι μη δεσμευτικό και να μην ε, και να μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις τοπικές δυναμικές. Για κάθε μακροπεριφέρεια απαιτείται ένα σχέδιο εκ των προτέρων σχεδιασμού, όπως είπαμε, το οποίο θα οργανώσει τη συνεισφορά των ενδιαφερομένων εταίρων θα σχεδιάσει του πρώτου ε, άξονε στρατηγική και θα καθορίσει επίση τι βάσει μια μελλοντική διακυβέρνηση. Σύμφωνα με τι αποφάσει του Συμβουλίου, η Επιτροπή αποτελεί τη φυσική διευθύνουσα αρχή μια τέτοια ενέργεια εκ των προτέρων σχεδιασμού. Πρέπει να διαθέτει του απαραίτητου ανθρώπινου και χρηματοδοτικού πόρου για τι σχετικέ επενδύσει, κυρίω βέβαια του ανθρώπινου πόρου. Τα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη προσπάθεια μακροπεριφερειακή συνεργασία προβλέπεται να αντιληφθούν στο πλαίσιο του στόχου 3 της πολιτικής συνοχής η Κομισιόν ανήγγειλε ότι θα αυξηθούν τα κονδύλια στο, για την περίοδο 2014-2020. Όλα αυτά μου φαίνεται ότι συνάδουν με την ανάπτυξη των μακροπεριφερειών. Η ενωτέρω χρηματοδοτική στήριξη πρέπει να λάβει τη μορφή πιστώσεων τεχνικής βοήθειας και για το στάδιο των προτέρων σχεδιασμού και για το στάδιο της υλοποίησης που θα προκύψει από το στάδιο των προτέρων σχεδιασμού. Τώρα, υπάρχουν, ε, ε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα, όπως είναι η, η συμπληρωματικότητα της χρηματοδότησης που πρέπει να γίνει ε, κριτήριο επιλογής υπέρ των μακροστρα, ε, περιφερειακών στρατηγικών όλων των σχεδίων που πραγματοποιούνται με βάση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ε, σε γενικές γραμμές αυτή είναι η εικόνα της μακροπεριφερειακής πολιτικής. Θα ήθελα να προσθέσω εν κατακλείδη ότι βρισκόμαστε σε μια ε, κρίσιμη σχετικά στιγμή. Δηλαδή έχουν ξεκινήσει ε, οι μακροπεριφέρειες υπάρχει μια νέα περίοδος προγραμματισμού η οποία ε, πρόκειται ε, να ξεκινήσει και πρέπει να σκεφτούμε τον τρόπο με τον οποίο οι θετικές αυτές επιπτώσεις θα ενταχθούν ίσως και καλύτερα στα μελλοντικά προγράμματα που, με τα οποία θα ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθώ στην σημασία της ε, μακροπεριφερειακής στρατηγικής στη Μεσόγειο. Ε, για σήμερα θα μείνω σε αυτό και αργότερα μπορεί να συζητηθεί το θέμα θα παραμείνω στα γενικά χαρακτηριστικά, είναι, που όμως δείχνουν αρκετά καλά το θέμα και για το λόγο για τον οποίο κατά τη γνώμη μου ε, η πρόθεση της ιδέας ότι μπορεί να υπάρχει στη Μεσόγειο μια μακροπεριφερειακή στρατηγική είναι σημαντική και γι' αυτό το λόγο έκανα αυτή την ε, προσπάθεια και διαβουλεύτηκα με τις περιφερειακές αρχές, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει μια διάθεση, για να μην πω προσδοκία, ε, για, προς αυτή την κατεύθυνση. Ποιες είναι οι τα βασικά αίτια. Ότι οι ακτές της Λεκάνης Μεσογείου ε, μοιράζονται το ίδιο φυσικό περιβάλλον, την ίδια ιστορική και πολιτιστική πραγματικότητα. Στην Νότια Ευρώπη Έχουμε εκατομμύρια κατοίκους που, είναι, που ζουν γύρω από τη Μεσόγειο. Υπάρχουν τεράστιες δυνατότητες, οι οποίες δεν θα μπορέσουν ποτέ να αξιοποιηθούν επαρκώς, χωρίς το συντονισμό και τη συνολική θεώρηση που επιτρέπει ο καθορισμός μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Δεύτερον, ότι στο χώρο αυτό που είναι ιδιαίτερα εκτενής τίθεται το θέμα του μακροπεριφερειακού μηχανισμού που θα πρέπει να προτιμηθεί. Στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχει Αδριατική και το Ιόνιο. Ε, θα κάνουμε ακρόαση εδώ για, με κάποιους από, τους, από τα στελέχη που θέλουν να προωθήσουν την περιοχή. Και υπάρχει και, αυτή η Ανατολική, και υπάρχει η Ανατολική Μεσόγειος. Θα πρέπει να εμβαθύνουμε το συντονισμό πριν επιλέξουμε αν θα κάνουμε μία ή δύο διαφορετικές μακροπεριφέρειες, μία της Δυτικής και μία της Ανατολικής Μεσογείου. Θα το δούμε αυτό. Πρέπει να εμβαθύνθει ο, συντον, ο, συντονισμός και η συνεργασία και θα το δούμε αυτό μέσω κάποιες ακρόασεις, να αποκτήσουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα από, για τις προσδοκίες και τις δυνατότητες. Τρίτο, η Μεσόγειος λόγω του κλίματός της του Μεσογειακού έχει περιφερειακού κότυπους κοινά προϊόντα, αγροτικά προϊόντα από την Ανατολή μέχρι τη Δύση και πολυμορφία παρόλα αυτά. Έχουν τα ίδια ε, ε, περιβαλλοντικά προβλήματα, ας πούμε τις πυρκαγιές και ε, υπάρχει επίσης αυτό το οικονομικό, σημαντικό οικονομικό πλεονέκτημα που, είναι ο που την κάνει πρώτο τουριστικό προορισμό και άρα είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν για τη διατήρηση και τη βελτίωση των προοπτικών αυτού του σημαντικού οικονομικού τομέα σε επίπεδο δυνατοτήτων πρέπει να τοποθετηθεί η θαλάσσια κυκλοφορία στο επίκεντρο μιας στρατηγικής για το τομέα των μεταφορών. Πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Οι θαλάσσιε οδοί πολύ συχνά αναφέρονται ε, από τους Ευρωπαίους οι αυτοκινητόδρομοι της ε, θάλασσας βλέπει κανείς ε, στο μυαλό του ένα αυτοκινητόδρομο, αλλά όταν μιλάμε για θάλασσα πρέπει να μιλάμε για τους θαλάσσιους δρόμους που είναι πολύ διαφοροποιημένοι και που επιτρέπουν ε, να, την ε, κοινωνία με απομακρυσμένες περιοχές και είναι σύνδεσμοι και ανακουφίζουν τα χερσαία δίκτυα. κυρίως το οδικό που προκαλεί μόλυνση και άλλες καταστροφές. Επιπλέον ένας ε, άλλος άξονας που είναι πραγματικά σημαντικός είναι το θέμα της ε, ε, ηλιακής ενέργειας. Και εδώ βλέπουμε στους στα κύματα των στόχων πώς μια μακροπεριφερειακή στρατηγική θα μπορούσε να, πλαισιώσει, να πλαισιωθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων. Η μεσογειακή βιοπικιλότητα επίσης είναι ένα σημαντικός παράγοντας, η οποία αποτελεί και πλούτο αλλά και ε, υφίσταται μεγάλες απειλές. Είναι μια κλειστή θάλασσα, μια ιδιαίτερα έντονη θαλάσσια κυκλοφορία και ε, το, η ποιότητα του περιβάλλοντος είναι σημαντική. Κυρίως ε, η, το, το περιβάλλον της θάλασσας αλλά και το παράκτιο περιβάλλον πρέπει λοιπόν να δει κανεί πώς θα μπορούσε να ενισχυθεί η συνεργασία Βορρά-Νότου μεταξύ των ε, ε, συλλογικών των αρχών των τοπικών αρχών. Αυτά είχα να πω όσον αφορά τώρα τα προσωπικά μου σχόλια. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να εντοπίσουμε τις ε, ε περιοχές της Ευρώπης όπου είναι ελλειπής η συνεργασία και υπάρχει έλλειμμα διασύνδεσης και συνεργασίας. Θεωρώ ότι η Μεσόγειος είναι ένα ε, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα ε, και με τη συνάδελφο μπορούμε να σας πούμε πόση ε, ε, έλλειψη υπάρχει συνεργασίας. Αυτά καταρχήν, κατόπιν. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το έλλειμμα σε αυτό το χώρο στη Μεσόγειο. Τώρα, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μεσόγειος είναι ε, ένας μεγάλος χώρος όπου κατοικούν 500 εκατομμύρια άτομα και δεν υπάρχει άλλη περιοχή κοντινή που να μπορεί να δεχτεί αυτούς τους ανθρώπους και κλείνοντας θα πω ότι θεωρώ ότι όλες αυτές οι δυνατότητες και όλες αυτές οι δυσκολίες οδηγούν τα κράτη και τις περιφέρειες της Ευρώπης που βρίσκονται στη Μεσόγειο να πρέπει να οφείλουν να ξεκινήσουν μια συνεργασία και για, το, για τον λόγο αυτό η μακροπεριφερειακή στρατηγική είναι ένας καλός χώρος. Η Πρόεδρος πρέπει... Έχουμε μόλις ένα τεταρτάκι και όταν είναι έτοιμο το σχέδιο κειμένου θα συνεχίσουμε. Τέλος Ιανουαρίου επομένω, παρακαλώ να είσαστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Ο Τόμας Ντόιτς είναι ο πρώτος που θέλει να λάβει το λόγο κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ναι, πιεζόμαστε ε, χρονικά, αλλά πρέπει να σας πω τρεις παρατηρήσεις. Πρώτα-πρώτα, να συγχαρώ τον κύριο Αλφονσί, γιατί δούλεψε σε βάθος και είναι πολύ αξιόλογο το έγγραφο το οποίο έχουμε για να συζητήσουμε. Επομένω και το έγγραφο ε, και όσο μας ε, εξήγησε ε, μας βοηθούν πάρα πολύ για να προχωρήσουμε. Έχω άλλες δύο παρατηρήσεις τώρα. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι συμφωνώ με τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Έτσι βοηθάτε πάρα πολύ η πολιτική της συνοχής για τις επόμενες δεκαετίες. είναι χρήσιμο και φιλόδοξο αυτό το εγχείρημα και βέβαια θα πρέπει να αξιολογείται και θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο με αυτή την έκθεση και την προετοιμασία αλλά και την ε, εφαρμογή και υλοποίηση της ε, στρατηγικής για Βαλτική και Δούναβη. Και είναι θέματα προτεραιότητας και τα δύο αυτά προγράμματα και τα δύο αυτά ε, οράματα. Δεν θα πρέπει ομένως να υποτιμήσουμε το γεγονός ότι εδώ έχουμε δύο μακροπεριφερειακές στρατηγικές. και να κάτσουμε και όσο γίνεται πιο προσεκτικά να κάνουμε μια αξιολόγηση. Και δεν πρέπει το ένα πρόγραμμα να είναι αιτία αναβολής του άλλου. Γιατί ό,τι κάναμε στο παρελθόν σε αυτό το μέτωπο μας ε, έχει δώσει πολύτιμη εμπειρία. Οπότε, θα πρέπει αντίθετα ό,τι κάνουμε σήμερα να βοηθάει για το ό,τι θα γίνει στο μέλλον. Επομένως, πρώτα-πρώτα θα πρέπει με κάποια κριτήρια ξεκάθαρα να αξιολογήσουμε την προπαρασκευή και την εκτέλεση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών μας. Τώρα, όσον αφορά τις μέλους στρατηγικές, έχουμε τις εξής ε, επιλογές. Τώρα βέβαια δεν λέω ότι πρέπει να αποφασίσουμε εδώ για τώρα. Όμως θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτές οι στατηγικές είναι τελείως διαφορετικές η μία από την άλλη. Πρώτα απ' όλα σε θεσμικό επίπεδο τα τρία θεσμικά όργανα προσπαθούμε να φτιάξουμε έναν χάρτη πορείας. που να επιδέχεται βέβαια κάποιες αλλαγές. Και να δούμε από πού θα ξεκινήσουμε για αυτές τις στρατηγικές. Άρα αυτό είναι προσέγγιση από πάνω προς κάτω. Από κορυφή προς βάση. Από την άλλη μεριά υπάρχει και η προσέγγιση αντίθετη από τη βάση προς την κορυφή και για τη Βαλτική και για τον Δούναβη. Μία ή η άλλη επιλογή. Φυσικά και υπάρχουν πολλά επέρ και πολλά κατά, αλλά δεν είναι δυνατόν να κάνουμε και τα δύο και τις δύο προσεγγίσεις. Εάν συνεχίσουμε με τις υπάρχουσες στρατηγικές, τότε δεν θα έχουμε και τίποτα σημαντικές αλλαγές. Εάν όμως διαλέξουμε την δεύτερη επιλογή, δηλαδή την προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, τότε νομίζω ότι τα πλεονεκτήματα θα είναι πολύ περισσότερα από τα μειονεκτήματα. Και γι' αυτό και εγώ είμαι υπεραυτής της δεύτερης επιλογής. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ θα χρησιμοποιήσω το χρόνο, τον λίγο που με έχει μείνει, για να σας πω ότι ο κύριος Αλφανσί Αν πέντε καφέ Για να δούμε. Το ότι θα να πρέπει να προσέξουμε εδώ δύο σημεία. Το είπε και ο κύριος Αλφονσέ, το ετώνησε. Πρώτα-πρώτα, όσον αφορά το πρώτο στοιχείο της μακροπεριφερειακής στρατηγικής, που είναι κάπως πιο πολύπλατο, θα πρέπει να δούμε ότι δεν θα πρέπει να υποκύψουμε στον πειρασμό του να ολιστήσουμε προς μια διακυβερνητική λύση. Γιατί η μακροπεριφερειακή στρατηγική πρέπει να μας οδηγήσει μακριά από αυτήν την κυβερνητική λογική. Να τον όσο γίνεται περισσότερο τον ε, ρόλο των περιφερειών και των τοπικών αρχών και των που περιφέρουν και των περιφερειακών αρχών. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μία μακροοικονομική οργάνωση. Γι' αυτό σύμφωνο επί του γεγονότος ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δύο διαστάσεις και να σκεφτούμε μία χαρτογράφηση για τις ε, μακροπεριφέρειες του μέλλοντος σε σχέση με το ιδιαίτερο θέμα της ε, Μεσογείου, θα επανέλθουμε σε αυτό, Νομίζω ότι από αυτή την άποψη, σε αυτή τη ζώνη, είναι δυνατόν να γίνει μια ιδιαίτερη εργασία, να ανακτήσουμε δηλαδή μια πρωτοβουλία σε σχέση με την Νότιο Ευρώπη, με το νότιο τμήμα της Ευρώπης και αναφέρουμε και στην άλλη όχθη της Μεσογείου, δηλαδή να έχουμε μια μεγαλύτερη παρέμβαση από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα και συμφωνώ με τις ε, δείξεις και τις υποδείξεις του Αλφόνση, ότι δηλαδή θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο η αναγκαιότητα μιας άλλης μακροπεριφέρειας που θα ήταν το Ιόνιο. Η Αδριατική και το Ιόνιο. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει μία ακρόαση με εκείνους που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρω ότι ως προς την Αδριατική και το Ιόνιο υπάρχει μία πρωτοβουλία όπου έγιναν πολλά προς αυτή την ε, κατεύθυνση και νομίζω ότι θα κατανοήσουμε σε ποιο σημείο ορίμανσης έχει φτάσει το σχέδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Οκατσίευσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Αλφόνση. Είμαι υπέρμαχος της, ε, του ορισμού νέων μακροπεριφερειών και συμφωνώ με πολλές δηλώσεις της έκθεσης. Νομίζω ότι έτσι θα επιλύσουμε οικονομικά και οικολογικά προβλήματα. Προωθούμε τη διασυνοριακή συνεργασία και ούτω καθεξής. Όμως σε αυτή την έκθεση δεν υπάρχει ένας σωστός, μια σωστή αποτίμηση και αξιολόγηση, δηλαδή να δούμε κατά πόσο οι μακροπεριφέρειες είναι ε, θετικές, ιδιαίτερα αυτές οι δύο. Δηλαδή, πώς, ε, ποιος είναι ο αντίκτυπος σε αυτή την περιφέρεια οι δράσεις των μακροπεριφερειών αφορούν τον ορισμό νέων μακροπεριφερειών. Επίσης θεωρώ ότι τα εδάφη όπου ορίζεται μία ε, μακροπεριφέρεια, θεωρώ ότι σε αυτή την περίπτωση όλοι οι δικαιούχοι ε, λαμβάνουν υπόψη τα τρία ναι. Δηλαδή, τη θέσπιση νέων κανόνων, μέσων και χρηματοδοτικών πόρων. Δεν μας είπε ο εισηγητής κατά πόσο πληρούνται αυτές οι προσδοκίες. Και δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη αυτών των μακροπεριφερειών. Εάν θεωρούμε ότι οι προϋπάρχουσες έχουν επιτύχει δεν θα πρέπει να αποκλείουμε νέες, γιατί όπου υπάρχει μια πρωτοβουλία από τα κάτω προς τα πάνω, θα πρέπει να ορίσουμε νέες μακροπεριφέρειες και νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μία άναντι προσέγγιση, συμφωνώ απόλυτα, όμως δεν αναφέρεται στην έκθεση κατά πόσο μπορούμε να ορίσουμε νέες μακροπεριφέρειες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Αλφονσί για το κείμενό του που είναι εξαιρετικό και συμφωνώ με τα συμπεράσματά του. Ε, στηρίζω τις πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις του και τρεις από αυτές πραγματικά μου φαίνονται ενδιαφέρουσες. Η δημιουργία ενός εκ των προτέρων σχεδιασμού που θα ε, βοηθήσει την εμβάθυνση, το, η του στόχου 3 για την τεχνική βοήθεια και η δημιουργία ενός χάρτη προβλέψεων ε, για τις μακροπεριφέρειες. Αντίθετα, το θέμα της επιλογής μιας ή δυο στρατηγικών, ανατολικής, δυτικής, ε, Μεσογείου κτλ. Αυτό πρέπει να συζητηθεί. Το θέμα αφορά και το μέγεθος της κλίμακας ε, πρέπει να επιμείνουμε στην ανάγκη συντονισμού με τα άλλα εφιστάμενα προγράμματα. Φερρυπίν, το Διεθνικό ΜΕΔ, ε, την ε, διασυνοριακή πολιτική γειτονία, η πρόταση της Ένωσης για τη Μεσόγειο και η Ένωση των εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρωμεσογείου. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε την πολιτισμική συνεργασία και τις ανταλλαγές σε θέματα παιδείας. Αυτές είναι πραγματικές προοπτικές ε, σε αυτό το χώρο. Τέλος, να υπενθυμίσουμε ότι οι τοπικές και περιφερειακές συνεργασίες που ε, καθημερινά δημιουργούνται μεταξύ Βορρά και Νότου επιτρέπουν να γίνει σημαντική πρόοδος για τον εκδημοκρατισμό των χωρών του Νότου όπως επίσης και οι μεγάλες διμερείς συμφωνίες που καμιά φορά δεν έχουν λειτουργικό περιεχόμενο. Ευχαριστώ κύριο Γκούτμαντς. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να προσθέσω κάποιες ε, απόψεις σχετικά. Πρώτον, όσον αφορά την ε, στρατηγική της Βαλτικής. Το πρώτο εδώ είναι ότι πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και οι γειτονικές χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα που προκύπτει. Για να πάει κανείς ε, στα, να βοηθήσει αυτά τα έργα χρειάζεται βοήθεια στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται στην περιοχή αυτή, οι οποίες αντιμετωπίζουν διαφορετικές συνθήκες και ε, που δημιουργούν προβλήματα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της περιοχής. Το δεύτερον, πρέπει να είμαστε πολύ ειλικρινείς. Υπάρχει μια αντίφαση μεταξύ των μακροπεριφερειών και των εθνικών κρατών αυτές οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές θα αρχίσουν να ζητούν επιπλέον πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πίτροπο Χακ έχει επισημάνει επανειλημμένως ότι αυτό δεν θα είναι εφικτό. Όμως πρέπει να πω και εγώ την αμαρτία μου. Έχω προτάσεις για την στρατηγική της Βαλτικής για το 2010-2011. Όχι πολύ μεγάλες, περίπου τάξος 20 εκατομμυρίων. Γιατί υπάρχουν κάποιες ανάγκες, πρακτικές ανάγκες, για την οργάνωση του όλου εγχειρήματο. Η απάντηση μέχρι τώρα είναι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Και θα πει σε απόθεμα γιατί δεν υπάρχουν έγγραφα που να αποτελέσουν την απαραίτητη βάση για τη χρηματοδότηση. Αυτοί οι οποίοι έχουν οργανώσει άλλες μακροπεριφέρειες ξέρουν ότι δεν θα υπάρχουν επιπλέον χρήματα για αυτές τις ανάγκες. Αν ναι, αν υπάρξουν πρέπει να το συμφωνήσουμε και να υποστηρίξουμε. Και δεύτερον, το θετικό εδώ είναι μόνο ένα. Αν δούμε τα ποσοστά απορρόφησης από τα εθνικά κράτη και θα σας παρουσιάσω το ποσοστό ε, απορρόφησης μέχρι 1η Δεκεμβρίου, σε 10 λεπτά όλα σε όλα τα μέλη θα το δώσω, πρέπει να πω ότι πολύ εύκολα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι το ποσοστό απορρόφησης είναι χαμηλότερο όπου συμμετέχουν διαφορε... όταν συμμετέχουν διαφορετικές χώρες, ακόμα και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δηλαδή, αν αυτές οι μακροπεριφέρειες ε, μπορέσουν με κάποιο τρόπο να επισπεύσουν το ρυθμό των διαφόρων χωρών για τη συμμετοχή τους σε κοινά έργα θα είναι θετικό. Και αυτός ίσως είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο έχει υποβληθεί αυτή η ιδέα και γι' αυτό πρέπει να την υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Σούτζε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εντάχει, θα ήθελα να συγχαρώ τον συνάδελφο Αλφονσί για την εξαιρετική αυτή εργασία, διότι μας παρουσιάζει ένα πλήρες κείμενο με τις κατάλληλες επιλογές εκεί όπου θα πρέπει να προβούμε σε εξειδικευμένες επιλογές, δηλαδή όταν θα πρέπει να ορίσουμε δύο μακροπεριφέρειες στα πλαίσια της Μεσογείου, γιατί μιλάμε για μια ευρύτατη ε, ζώνη από γεωγραφικής πλευράς, η οποία έχει κοινά προβλήματα. Νομίζω λοιπόν ότι πληρούνται όλοι οι όροι για να προχωρήσουμε σε αυτή τη βάση και νομίζω ότι επίσης τονίζεται η δύναμη της μακροπεριφέρειας στη συνέργεια αυτή που δημιουργείται. Με βάση δηλαδή μια κοινή συλλογιστική για να έχουμε μια ε, μεγαλύτερη εξέλιξη για αυτή την περιφέρεια. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να πει κάτι ο Φρανσουά. Έχει ένα λεπτό. Μέσα σε ένα λεπτό θα πω ότι ευχαριστώ όλους όσοι διάβασαν προσεκτικά το κείμενό μου. Ευχαριστώ για τα, για τα σχόλια και τις προτάσεις τους. Θέλω απλώ να πω ότι ετέθη ένα θέμα για το UPM, ένα σημαντικό, ότι είχα πάει σε ένα φόρουμ ε, στην Σικελία, από την περιφέρεια της Σικελίας είχε οργανωθεί. Στην, στην αρχή δεν ενδιαφέρθηκαν, μετά εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για, το, για τη μακροπεριφέρεια, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι ίσως η καλύτερη βάση για να προχωρήσει η ευρωμεσογειακή στρατηγική και στις 27 Ιανουαρίου θα πάω στη Βαρκελόνη και θέλω να πω στους και όλους τους και στους ενδιαφερόμενους συνάδελφους ότι αν θέλουν να με συνοδεύσουν στην αντιπροσωπεία αυτή είναι σαφώς ευπρόσδεκτοι και βεβαίως θα τους ενημερώνω τακτικά κάθε φορά που γίνεται μια τέτοια συνάντηση. Και για να κλείσω και να μην παραβώ το χρόνο μου, οι επαφές που είχαμε και που θα έχουμε από αυτές του Ιανουαρίου ε, μου ζητούν κάθε φορά να γίνει μια μικρή, μια μίνι ακρόαση στα πλαίσια της Επιτροπής μας, ώστε η Επιτροπή να μπορέσει να ακούσει τους συνομιλητές που έχω συναντήσει και οι οποίοι συχνά πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό το έργο το οποίο τους παρουσιάζω. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, είναι φοβερά φορτωμένη η ημερήσια διάταξη του Ιανουαρίου, αλλά θα δούμε τι θα μπορεί να γίνει. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Το σχέδιό μας είναι τον Ιανουάριο να ακούσουμε την, ε, το σχέδιο έκθεσης και να συζητηθεί στην ε, Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Περνάμε σε ένα χθεσινό θέμα που δεν μπόρεσε να συζητηθεί, το ε, η εξέταση για το σχέδιο γνωμοδότηση στο μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και υπηρεσιών. Έχουμε μόνο 20 λεπτά. Σας παρακαλώ να είστε όσο το δυνατόν πιο σύντομο, κύριε Ούτζα. Ευχαριστώ. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Όπως και το κείμενο το οποίο σας υπέβαλα. Θα ήθελα να κάνω δύο ανακοινώσεις πρακτικής υφής. Ότι δυστυχώς η υποβολή τροπολογιών, η προθεσμία είναι πολύ κοντινή. Ορίστηκε για αύριο, για οργανωτικούς λόγους και για να εξετάσει το κείμενο και η Επιτροπή Τραν. Επειδή λοιπόν Έχουμε και τη, τα Χριστούγεννα δεν, που μεσολαβούν δεν μπορούσαν να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό θα ήθελα να ε, συλλέξω όλες τις ε, παρατηρήσεις και να συντάξουμε με τα γενέστερα συγκεκριμένες τροπολογίες συμβιβασμού. Το ε, κείμενο αφορά 7 παραγράφους που για, εσωτερικές, για εσωτερικούς λόγους θα πρέπει να τηρήσει αυτή τη δομή. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Χρειάστηκε να ε, κάνουμε περικοπές και να διαγράψουμε και λέξεις. Γι' αυτό έκρινα σκόπιμο να σας μιλήσω για ορισμένες προτεραιότητες και στη συνέχεια θα μπορέσουμε να διευρύνουμε το κείμενο υπό μορφή τροπολογιών. Έτσι θα έχουμε περισσότερο χώρο και θα, θα μπορέσουμε να ενσωματώσουμε και άλλα θέματα επειδή θα πρέπει να κάνουμε υποδείξει στην Επιτροπή Τραν για το μέλλον των ε, αεροπορικών υπηρεσιών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έπρεπε να δούμε ποια είναι τα περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία ορίζουν την εδαφική συνοχή, παράγραφος 1. Ποιος είναι ο ρόλος των περιφερειακών αεροδρομίων για να δημιουργήσουν και απασχόληση, παράγραφοι 2 και 3. Ε, τρίτον, παράγραφος 4. Το θέμα του περιβάλλοντος και ο διατροπικός χαρακτήρας, παράγραφος 5 για να ορίσουμε και τα χρηματοοικονομικά μέσα. Ως προς το πρώτο θέμα, έκρινα ότι, και κρίνουμε όλοι ότι τα περιφερειακά αεροδρομία διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για την πολιτική συνοχή της Ευρώπης για να συνδέσουν όλους τους τομείς και περιφέρειες, για να συνδέσουν τις απομακρυσμένες περιοχές, νησιά και ούτω καθεξής για να μπορέσουμε να συνδέσουμε τις ευρωπαϊκές περιφέρειες θα πρέπει να ορίσουμε ένα πλαίσιο ε, αναφοράς το οποίο να είναι επαρκές για τις υποχρεώσεις του δημόσιου τομέα. Η δεύτερη και τρίτη παράγραφος ορίζουν την ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων έτσι ώστε να προωθήσουμε και τον τουρισμό που είναι ύψης της σημασίας για πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες και να λειτουργήσει ως καταλήτης, να λειτουργήσουν ως καταλήτης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα στις μεονεκτούσες περιοχές όπου θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, εκεί όπου η ανεργία είναι υψηλή. Η ιδέα του πρασινίσματος ορίζει την τέταρτη παράγραφο για να λάβουμε υπόψη μετεωρολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες τη στιγμή που εντοπίζουμε τα αεροδρόμια αυτά. Η πέμπτη παράγραφος μιλά για περιφερειακή προσβασιμότητα γιατί αυτό που μας ενδιαφέρουν είναι και οι διατροπικές συνδέσεις, δηλαδή και οι σιδηροδρομικές μεταφορές, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τρένα υψηλής ταχύτητας. Πρόκειται για πρωταγωνιστικούς τομείς για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διατροπική σύνδεση λαμβάνει υπόψη το συνδυασμό σιδηροδρόμων και αεροδρομίων. Και τέλος, συνάδελφοι, έκρινα σκόπιμο να ε, γίνει μία επαρκής αναφορά στην χρηματοοικονομική υποστήριξη των αεροδρομίων αυτών μέσα στα πλαίσια των δικτύων TEN, καθώς ε, και ένα θέμα εδαφικού προγραμματισμού όπου θα συνδράμουν και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές σε... και θα συνεργάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ωραία λέει η Πρόεδρος και ο Ισκιώδης τώρα, ε, Γιώσεφ Μάτουλα. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχολεία. με σκιώδης από το ΕΛΚ. Θα πρέπει να δούμε τις ε, συμβατικές, ε, τις εταιρικές συμβάσεις που θα πρέπει να ενταχθούν στη στρατηγική περιφερειακής ε, ανάπτυξης και θα πρέπει να αναφέρονται στις μελλοντικές εταιρικές συμβάσεις. Δεύτερον, η διευκόλυνση σύνδεσης η πανευρωπαϊκή, ο πανευρωπαϊκός μεθοδολογικός προγραμματισμός, ο οποίος θα πρέπει να λάβει υπόψη τις δυνατότητες που ε, δίδουν τα περιφερειακά αεροδρόμια στα, ως προς τις κεντρικές διασυνδέσεις. Ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη, τα περιφερειακά αεροδρόμια ε, δημιουργούν κινητικότητα και συνδεσιμότητα μεταξύ περιφερειών για να προωθήσουμε και τουριστικές δραστηριότητες. Τέταρτον, ε, επανακίνηση των περιφερειακών αεροδρομίων για χαμηλότερες δαπάνες και άμεσα πλεονεκτήματα για να βοηθήσουμε στην αποσυμφόρηση των μεγάλων αεροδρομίων. Παράλληλα, συνεισφέρουν στην διαφοροποίηση των, ε, της ε, διασυνδεσιμότητας. Και το πέμπτο σημείο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα γειτονικά περιφερειακά αεροδρόμια και εδώ θα μπορούσαμε να βρούμε ε, διατροπικές συνδέσεις, δημιουργώντας απασχόληση, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα και την κινητικότητα της περιφέρειας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιώσεφ. Ο κύριος Καρόνα. Ε, Νομίζω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ σημαντική παρά το γεγονός ότι είναι μία σύντομη έκθεση, γιατί τα μικρά περιφερειακά αεροδρόμια τα δέκα τελευταία χρόνια γνώρισαν μεγάλη ανάπτυξη. Είτε ως προς τον αριθμό των επιβατών, που αυξήθηκε πάρα πολύ, είτε ως προς ε, την ανάπτυξη των υποδομών. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία σε αυτά τα αεροδρόμια. Καταρχήν, βλέπουμε ότι υπάρχει μια συγκέντρωση περιφερειακών αεροδρομίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία δεν ακολουθεί ε, έναν μια ορθολογική δομή και πολλές φορές επικρατεί τοπικισμός που δεν βοηθά στη συμπλήρωση του συστήματος. Ένα άλλο στοιχείο έχει ως εξής. Αν από τη μία πλευρά υπήρχε μεγάλη ανάπτυξη ορισμένων περιφερειακών αεροδρομίων, και αυτό αφορά τις εταιρείε low cost, υπήρξε μία αύξηση της απασχόλησης αλλά παράλληλα δυστυχώς δεν πληρούνται οι σωστοί όροι εργασίας των εργαζομένων. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Τέλος, και το ανέφερε ήδη ο εισηγητής, η πολιτική συνοχής μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα ε, ως προς τις διατροπικές συνδέσεις και από αυτή την άποψη θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον συνάδελφο κύριο Γκίας για τη σύνταξη αυτού του σχεδίου γνωμοδότησης της Επιτροπής μας και να κάνω κάποιες επισημάνσεις σχετικά με το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων και τις εναέριες υπηρεσίες στον χώρο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως πράσινοι εκτιμούμε ότι δεν είναι η αναγκαία η κατασκευή περισσότερων αεροδρομίων παρά μόνο σε υπερβολικά απομακρυσμένες περιοχές, εκεί όπου η σύνδεση με την κυρίως χώρα είναι προβληματική. Επιπλέον, ε, τα αεροδρόμια θα πρέπει να έχουν καλή σύνδεση με μέσα μαζικής μεταφοράς, σωστά λέει η έκθεση, και τονίζουμε τη σημασία των συνδυασμένων μεταφορών και θέτω εδώ, για παράδειγμα, το ζήτημα της δημιουργίας σιδηροδρόμου στην Κρήτη και στην Κύπρο που δεν υπάρχει καμιά ε, σιδηροδρομική υποδομή. Ε, δεν είμαστε υπέρ της ιδέας των περιφερειακών ε, αεροδρομίων όπως έχει επικρατήσει και επιδοτούνται ε, συνήθως από τα κράτη. Το μικρό και περιφερειακό αεροδρόμιο συχνά δεν έχει το απαραίτητο κέρδος και ως αποτέλεσμα έχουμε οι αεροπορικές εταιρείες να φεύγουν από τα τοπικά αεροδρόμια και να κλείνουν. Ε, υπάρχουν ε, οι εταιρείες, οι αεροπορικές χαμηλού κόστους που δεν πληρώνουν ε, φόρους αεροδρομίου με αποτέλεσμα οι περιφέρειες να μην έχουν έσοδα και τα περιφερειακά αεροδρόμια να αποτελούν κάποιες φορές έναν τομέα χωρίς προοπτική. Οι συνθήκες εργασίας δεν είναι ιδανικέ για τους περισσότερους που απασχολούνται σε τέτοια αεροδρόμια και οι συμβάσεις προέρχονται από χώρες το, ε, όπου προέρχονται οι αεροπορικές εταιρείες. Ε, έτσι τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία σχέση με τις τοπικές συμβάσεις και τους κανονισμούς. Και μπορεί να καταλάβει κανείς τις επιπτώσεις και για τους εργαζόμενους και για τις ε, περιοχές. Στην Ελλάδα ε, μπορώ να πω ότι η κατάσταση ε, στα νησιά ε, φανερώνει ότι δεν χρειάζονται άλλα αεροδρόμια. Πολλά είναι αρκετά μικρά ούτως ή, άλλο, για να δεχθούν αεροδρόμια και πολύ συχνά η κατασκευή τους είναι επιβαρυντική και βλαπτική για το περιβάλλον και επίσης ανταγωνιστική με τη γεωργία και την κατοικία αλλά και τις τουριστικές ε, υποδομές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στην προώθηση των ε, περιφερειακών τέτοιου είδους αεροδρομίων. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, Ευχαριστώ η Μαρίτα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο που έκανε αυτή την πολύ συνοπτική έκθεση με τις λίγες παραγράφους. Δύο-τρία σημαντικά σημεία για τον ε, θετικό ρόλο των περιφερειακών ε, αεροδρομίων στην περιφερειακή ανάπτυξη. Η σημασία για τον τουρισμό και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, η ιδέα της ενσωμάτωσης των ε, περιφερειακών αεροδρομίων στην περιφερειακή χώρα στο περιφερειακό χωροταξικό σχεδιασμό και επίσης τη δυνατότητα να μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής και από το ΦΕΝΤΕΡ. Αλλά θέλω να αναφερθώ στη δυνατότητα της διαμεθοριακής συνεργασίας, όχι μόνο για να ε, χρησιμοποιούνται από κοινού εξοπλισμός, αλλά και για την ε, κοινή χρήση των δικτύων των οδών κλπ. Αυτό είναι κάτι που πρέπει και να το αναφέρουμε και να το διερευνήσουμε. Ευχαριστώ η Ελίζα Σρέτερ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα απλώς να υπογραμμίσω αυτό που είπε η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών σε σχέση με αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα του των όρων εργασίας που προσφέρουν αυτές οι αεροπορικές εταιρείες. Το βλέπουμε αυτό παντού. Εμένα στη χώρα μου προσπαθήσαμε να, να το κάνουμε αυτό και διαπιστώσαμε ότι είναι χαμηλός ο αριθμός. Χαμηλό το επίπεδο του ανταγωνισμού και δεν έχουν προκύψει πολλά ωφέλη. Πρέπει να πούμε τι έγινε. Ίσως τα βγάζουν πέρα στην αρχή τα αεροδρόμια, αλλά όταν έχουν να αντιμετωπίσουν το πραγματικό κόστος αργότερα, ε, πτωχεύουν και έχουν διαρκώς ε, ε, ανάγκη από ενισχύσεις και άλλες ενισχύσεις και άλλες ενισχύσεις. Το έχουμε αυτό το πρόβλημα στη Γερμανία και διαρωτώ με αν πραγματικά αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Δηλαδή, αν σε αυτό ε, Προσθεθεί το γεγονό ότι ω Ευρώπη έχουμε δεσμευτεί για την προστασία του κλίματο, θα πρέπει κανεί στα σοβαρά να διαρωτηθεί μήπω δεν θα έπρεπε να αναθεωρηθεί αυτού του είδους η ενίσχυση και να προσπαθήσουμε να βρούμε άλλες εναλλακτικέ λύσεις ε, προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Μια ε, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με τη δημιουργία πραγματικών θέσεων εργασίας ε, βάσει των οποίων θα μπορεί κανείς να ζήσει και με το σεβασμό στο περιβάλλον που θα επιτρέψει να επιβιώσουν στο μέλλον οι γενιές, οι ερχόμενες γενιές. Αυτά είναι τα θέματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, να σκεφτούμε το κλίμα και να σκεφτούμε το γεγονός ότι θέλουμε να είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο για να ξεκινήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση και έχουμε ανάγκη να το κάνουμε. Για όλους αυτούς τους λόγους διερωτώ με σοβαρά αν μπορούμε να ε, στείλουμε μια τέτοια γνωμοδότηση. Διερωτώ να το μήπως θα πρέπει να το προσεγγίσουμε υπό το πρίσμα των συνδυασμένων μεταφορών της κοινωνικής διάστασης και της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Για μένα η γνωμοδότηση αυτή πραγματικά θα πρέπει να ασχοληθεί με το αν και κατά πόσον στο μέλλον θα έχουμε ανάγκη από τέτοιου είδους αεροδρόμια και αν πρέπει να τα ενισχύσουμε. Ευχαριστώ. Πρέπει να εξηγήσω, λέει η Πρόεδρος, γιατί υπάρχει αυτή η τόσο σύντομη ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Αν θέλουμε να φτάσουν στην Επιτροπή Μεταφορών για, για την ε, ψηφοφορία και αφού η ψηφοφορία θα γίνει το Φεβρουάριο, Πρέπει η γνωμοδότηση να είναι έτοιμη στις 25 Ιανουαρίου και τώρα επειδή υπάρχει η δυσκολία των γιορτών των Χριστουγέννων και το θέμα της μετάφρασης δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα παρά να θέσουμε αυτή την ε, προθεσμία αύριο. Επίσης, έχουμε στείλει εδώ και δύο εβδομάδες τη γνωμοδότηση σε όλους τους σκιώδεις για να έχουν τον επαρκή χρόνο να την ε, επεξεργαστούν. Ελπίζω οι συνάδελφοι να χρησιμοποίησαν αυτό το χρόνο και ότι η αυριανή προθεσμία δεν θα αποτελέσει πρόβλημα για κανέναν. Ε, και ένα λεπτό ακόμα στον Τζαν Μαρία για να πει ε, τις απόψεις του. Όλα τα σχόλια είναι ποιοτικά σχόλια και θα ενταχθούν στο κείμενο, το οποίο είναι πολύ σύντομο, όπως γνωρίζετε, για λόγους ε, αναγκαιότητας. Και εγώ θα υποβάλω ορισμένες τροπολογίες, έτσι ώστε να διευρύνω κάπως το κείμενο. Βεβαίως, θα λάβουμε υπόψη τις κεντρικές ε, περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δούμε και τους όρους εργασίας των εργαζομένων, η σύνδεση με άλλα μέσα μεταφοράς, ο νησιωτικός χαρακτήρας απομακρυσμένων περιοχών. Όλα αυτά θα ενσωματωθούν. Θα ήθελα να πω όμως ε, το εξής και μόνο στους συναδέλφους, γιατί είμαι σκιώδης και στην Τραν, όπως ξέρετε, και η ΤΡΑΝ δεν είναι σαφής ως προς τον ορισμό του περιφερειακού αεροδρομίου. Δηλαδή θεωρεί ότι είναι περιφερειακά αεροδρόμια ε, όλα τα αεροδρόμια της Ευρώπης που δεν ε, βρίσκονται στην πρωτεύουσα. Δηλαδή η Φραγκφούρτη με αυτή τη λογική είναι περιφερειακό αεροδρόμιο, όπως καταλαβαίνετε. Άρα θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα το θέμα είναι ένα ουσιαστικό θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Θα προωθήσω αυτές τις πληροφορίες και στους συναδέλφους όταν και όπως ανακύπτουν. Ευχαριστώ. Κλείνουμε αυτό το θέμα αγαπητοί συνάδελφοι και θα ήθελα να σας πω ότι η προθεσμία είναι αύριο 21 Δεκεμβρίου 12 το μεσημέρι. Ε, για όσους θέλουν να υποβάλουν τροπολογίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα ήθελα να επανέλθω σε ένα σημείο που ανέφερα χτες για αυτούς που δεν ήταν παρόντες. Ξέρετε, με τη Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο έχουμε ε, την ε, ανάπτυξη ενός κεντρικού σημείου ο κύριος Μπούτζαχερ προήχθη και ίσως το θέμα αυτό απασχολεί την Τσεχία, τη Σλοβενία, την Αυστρία. Ε, ε είσαστε και εδώ, μπορείτε να μας ε, πείτε δύο λόγια αν θέλετε, επί την προαγωγή. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κυρία Χίμπνερ για την ε, ευκαιρία που μου δίνετε να αποχαιρετήσω. Μάλλον καλύτερα να πούμε στο επανειδήν, ρεβουάρ στα γαλλικά, κάτι το οποίο είναι πιο θετικό. Όντως, πήρα προαγωγή. Οπότε, αυτό είναι το κάλεσμα του καθήκοντος. Οπότε, θα πρέπει να σας ε, ομολογήσω και να παραδεχτώ ότι πάρα πολύ ε, ικανοποιητικά ήταν τα, όσα γίνανε για αυτές τις δύο τροπικές ε, προτάσεις ε, και τώρα επιτέλους έχουμε την ε, θέση σε ισχύ της πιο πρόσφατης τροποποίησης και τροποποιημένης εκδοχής τέλος πάντων του νομοθετήματος αυτού. Είμαι βέβαιος ότι θα ξαναέρθω, θα με ξανακαλέσετε διότι θα προκύψουν και άλλα θέματα σε σχέση με τις τωρινές μου αρμοδιότητες αυτές τις χώρες τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και στα γερμανικά να ευχηθώ σε όλους καλά Χριστούγεννα, καλή χρονιά και ήταν πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συνεργασία μας, ιδίως δύο τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ. Γεια σας. Αυτό σημαίνει ότι βοηθάει, βοηθάει στη σταδιοδρομία το να συνεργάζεται κανείς με το κοινοβούλιο, άρα αυτό να το έχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι κατά νου. Τώρα, θα θυμάστε οι παλαιότερο τον Φαμπρίτσιο Μπάρκα. Τώρα είναι υπουργό της νέας Ιταλικής κυβέρνησης. Και το χαρτοφυλάκιό του καλύπτει πάρα πολλά θέματα σε σχέση με ε, την περιφερειακή ανάπτυξη και την περιφερειακή συνοχή. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτή η πρόκληση που να αντιμετωπίσει. Ευχαριστούμε που ήρθες να μας δεις. Αλλά έχουμε και την κυρία Ντελούκα που ανέκαθεν συμμετέσχε στα θέματα ε, πολιτικής συνοχής στις ιταλικές ε, κυβερνήσεις. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Μπάρκα. Ναι, τώρα ήρθα υπό άλλη ιδιότητα και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τώρα να σας τα πω αγγλικά και συμπαθάτε με, συμπατριώτες. Και στις 15 Δεκεμβρίου, από τρεις μέρες, επί... εξεργαστήκαμε αυτό το σχέδιο δράσης, το ώστε να αξιοποιήσουμε 3,1 δις για τις προτεραιότητές μας, δηλαδή την ε, ψηφιακή ατζέντα, τα ψηφιακά θέματα, παιδεία, σιδηρόδρομοι και κάποια λίγα από αυτά τα χρήματα για τα πρόσωπα με ειδικέ ανάγκες και τα μισά από αυτά τα χρήματα θα αφορούν τα περιφερειακά προγράμματα και προήλθαν από την αύξηση του συντελεστή συγχρηματοδότηση για την Ιταλία. Ήμασταν στο 50% του υψηλότερου δυνατών. Τώρα 1,5 δις έχουν εξοικονομηθεί από την προσαρμογή αυτού του ποσοστού και όλα θα πάνε στους δρόμους Σύμβουλο και η Επιτροπή είπαν και επεκύρωσαν αυτή την απόφαση στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφής. Και οι επιπτώσεις θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικέ και γι' αυτό και χαίρομαι που βρίσκομαι να το συζητήσουμε γιατί έτσι θα δείτε πώς βλέπει η νέα μα κυβέρνηση το πώς μπορούμε ταυτόχρονα να επιταχύνουμε τις δαπάνε και ταυτόχρονα να τις κάνουμε πιο αποτελεσματικές από πλευρά αναπτυξιακή. Όλα αυτά αφορούν την πολιτική συνοχή, όλα αυτά προβλέπονται από το σχέδιο κανονισμού και όλα αυτά νομίζω ότι ε, πήγαν πάρα πολύ καλά λόγω του εξαιρέτου έργου της Πολωνικής Προεδρίας. Κυρία Χίμνερ, το ότι βρίσκομαι εδώ αποδεικνύει το πόσο ε, σημαντικό θεωρούμε ότι είναι το να έρχονται εδώ εκπρόσωποι των μελών για να τα συζητούμε. και έτσι να διαπιστώνεται η αποτελεσματική απορρόφηση αυτών των κονδυλίων. Άρα, θα πρέπει να διαπιστωθεί ότι η Ιταλία βρίσκεται πάρα πολύ πίσω όσον αφορά την απορρόφηση των κοινωνικών κονδυλίων. Είμαστε στην πρώτη τελευταία θέση της σχετικής κατάταξης και κυρίως η Νότια Ιταλία. Είχαμε σύγκληση 12% δηλαδή το μισό του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, δεν ήταν πάντοτε έτσι τα πράγματα. Τα πράγματα έχουν επιθυμωθεί στην Ιταλία. Καλά, όλα τα κράτη-μέλη ε, πάνε χειρότερα όσον αφορά την απορρόφηση των κονδυλίων, αλλά εμείς, εμείς, αν κανείς συγκρίνει τα σχετικά στοιχεία, θα δείτε ότι έχουμε κατρακυλήσει κατά εννέα μονάδες. Τρίτον, και αυτά είναι τα καλά μαντάτα μέσα στο δυσάρεστο ε, αυτό το έχουμε ακόμα και στις περιοχές σύγκλησης, έχουμε κάποιες περιοχές σαν την Μπαζιλικάτα που βρίσκονται κοντά στον μέσο όρο, αλλά ακόμα δεν έχουν πιάσει το 10%. Και έχουμε εθνικά προγράμματα όπως το πρόγραμμα παιδείας που πάει στο 40% αφορά τις δαπάνες, επομένως αυτά σαν αφετηρία. Τώρα, τέσσερις λόγοι γιατί πήγαμε σε αυτήν την κατάσταση. Είναι δύο παλιά προβλήματα και δύο επιπρόσθετα. Η κατάτμιση της παρέμβασης, δεύτερον, η ανεπαρκής εστίασε στα αποτελέσματα. σε σχέση με τις επιδόσεις στην ευημερία και το ιδιωτικό επίπεδο. Δεν το προσέξαμε αρκετά. Και, όπως είπαμε και στο Κοινοβούλιο πριν από δύο μέρες, ότι έχουμε επιδείνωση όσον αφορά την εθνική διακυβέρνηση, ιδίω όσον αφορά κάποια βασικά σημεία σύγχυση μεταξύ αποκέντρωσης και συρρήγνωσης του ρόλου της κυβέρνησης. Σε σχέση με την εποπτεία και τον εντοπισμό των προβλημάτων. Και είπαμε ότι το ένα συνετέλεσε μαζί με το άλλο πρόβλημα. Και επίση υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αβεβαιότητα, και καταλαβαίνετε τι λέω, ότι αυτή η αβεβαιότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τις περικοπές αλλά και το ότι θα ακολουθήσουν και άλλες περικοπές και επίσης το ότι υπάρχει ένα εσωτερικό σύμφωνο σταθερότητας για την Ιταλία έχει λάβει ομοσπονδιακή κατεύθυνση. Και επομένως έχουμε την συγχρηματοδότηση σε σχέση με την συνεργασία μας με τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτή ήταν η λόγη, αυτή ήταν η διάγνωση και η θεραπεία θα είναι ως εξής. Έχουμε τι τέσσερι προτεραιότητε όπου θα κατευθύνουν ε, αυτά τα χρήματα που είπαμε πριν. επίση έχουμε το ότι θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μας στα αποτελέσματα και έχω ετοιμάσει για εσά ένα σύντομο σημείο μια σελίδα το οποίο θα σα το διαβιβάσω και είναι αυτό η σύνοψη των σα είπα, Επομένω, εστιασμό στα αποτελέσματα δηλαδή. Κάνουμε αυτά τα οποία λέει ο κανονισμό. Πόσα χρήματα έχουμε, τι θα κάνουμε και τι στόχους έχουμε θέσει. Και ξεκινούμε από τους στόχους. Ποια από τα προβλήματα της Νότιας Ιταλίας θα έχουμε θέσει ως στόχους μέχρι τις 31 πρώτη. κατόπιν τι θα κάνουμε για να πετύχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα και μετά πόσα χρήματα θα δαπανίσουμε και άρα κατά κάποιο τρόπο αντιστρέφουμε την ε, στρατηγική. Τρίτον, θα θέλουμε να υπάρχει χρηματοδοτική βεβαιότητα η οποία θα προκύψει από την κυβέρνηση λόγω αυτή, αυτών, αυτών των λιγμών, αυτή της ε, σκληρής τακτικής, αλλά έτσι θα αποφύγουμε άλλες ε, τέτοιες πολιτικές και θα έχουμε λιγότερη αβεβαιότητα και επίσης έχουμε και την απάντηση σε αυτή την επιστολή που πήραμε από τους ε, συναρμόδιους επιτρόπους του Γεωργίου Γεωργάν που είπαν ε, ναι να κάνετε αυτό το σύμφωνο σταθερότητα, αλλά να μην οδηγήσετε τι περιφέρειες στο να μην δαπανώνουν αυτά που πρέπει να μην απορροφούν. Και τώρα με νόμο δεν θα περιορίζονται όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση οι περιφέρειες της χώρας. Τέταρτον, κινητοποίηση των εθνικών κέντρων το Υπουργείο Παιδείας τώρα παρεμβαίνει στα λειτουργικά προγράμματα για την εκτελεσή τους. Εξασφαλίζει την εκτέλεση των προγραμμάτων στα σχολεία παντού όπου χρειάζεται, ούτως ώστε να είναι αποτελεσματική η εκτέλεση των προγραμμάτων. Τώρα, ποιες είναι συνέπειες στην ανάπτυξη. Υπάρχουν κάποιες ε, άμεσες συνέπειες. Δεν ξέρω αν θα άρεσαν αυτά στον Κέινς αλλά πάντως υπάρχουν κάποια βραχυπρόθεσμα που δεν πρέπει να γνωρίσουμε. Και θα πρέπει να στεναχωριόμαστε ότι αυτά τα οποία κάνουμε θα έχουν κάποιες συνέπειες όπως το ότι θα ανέβει το εισόδημα των διδασκόντων στην Ιταλία που δεν αμείβονται αρκετά όπως λέει ο ΣΑ. Άρα θα πάνε κάποια χρήματα στην τσέπη αυτών που δουλεύουν. Και επίσης και για τους μη προνομιούχους εργαζομένους έχουμε ε, κάποια ωφέλη για γυναίκες, για κάποιους που είναι πάνω από 40, για κάποιους που έχουν πάνω από 24 χρόνια δουλειάς και το πιο σημαντικό είναι βέβαια ότι έχουμε και κάποια μέσα αποτελέσματα αυτό το οποίο έχουμε θέσει ως στόχο, δηλαδή θέλουμε το κοινωνικό συμβόλαιο του Νότου με το κράτος να γραφτεί από την αρχή. Να ξεκαθαριστεί τι προσδοκάται να κάνει το κράτος για αυτούς που κάθε μέρα θέλουν να πάνε στη δουλειά τους στο σχολείο. Πολύ σημαντικά αυτά και μακρόπνα. Επίσης, τελευταίο σημείο είναι το τι περιμένουμε, τι προβλέπουμε όσον αφορά αυτές τις αλλαγές. μέχρι το 2014 ελπίζουμε τα εξή να έχουν προκύψει αυτά τα οποία προανέφερα ότι αντιστρέψαμε την στρατηγική και τα αποτελέσματα στην ευημερία και στη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου είναι οι δείκτες, τα κριτήρια, το επίκεντρο των πολιτικών μας και επίσης λέμε με τι δράσεις θα πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα με διαφάνεια και εξηγούμε γιατί πιστεύουμε ότι αυτές οι δράσεις θα πετύχουν τα αποτελέσματα. Τα είπαμε και στο Συμβούλιο ότι αυτά τα λειτουργικά προγράμματα θα πρέπει να πλουστευτούν κατά πολύ σε σχέση με αυτό το οποίο, με αυτό τον άξονα. Αποτελέσματα, δράσεις και το πώς θα λειτουργήσουν οι δράσεις για αυτά τα αποτελέσματα. Επίσης, τρίτον και πολύ σημαντικό, η σύνδεση με τις τομιακές πολιτικές. Και θα πρέπει αυτό να αφορά και τις περιφερειακές πολιτικές. Σε κάποια κράτη-μέλη αυτά τα κονδύλια, το οποίο ισχύει και την Ιταλία, έχουμε απομόνωση, κατάθμιση, αποσύνδεση αυτών των πολιτικών. Και αυτό έχει να κάνει και με πάρα πολύ σημαντικά κονδύλια τα οποία πάνε στην παιδεία. Άρα θέλουμε με αυτό το δις το οποίο θα πάει στην παιδεία θέλουμε να σχετιστεί και με το τι κάνουμε στις τομιακές πολιτικές. Άρα θα πρέπει η τομιακή πολιτική για τον Νότο να προσαρμοστεί σε αυτά τα οποία θέλουμε για την περιφερειακή πολιτική. Τελευταίο τώρα, εν κατακλείδη. Όπως τα είπε και ο πρόεδρος Μόντι, θέλουμε να έχουμε αναβαθμισμένη συνεργασία ισχυμένη συνεργασία μεταξύ τη κυβέρνηση και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρω ότι εσεί όταν ε, λέτε ισχυμένη συνεργασία εννοείτε κάτι άλλο, αλλά έχουμε μια ομάδα δράση, τη οποία ε, προεδρεύει η κυρία Ντελούκα, εδώ που στα αριστερά μου, και έχουμε και αντιπρόεδρο, έναν διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που για μα είναι πάρα πολύ σημαντική κίνηση. ε, επικουρικότητα σε βάθος το όνομα αυτό ο πρόεδρος ότι... Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Συζήτηση τώρα. Κωνσταντσα Κρέλ είναι η πρώτη που έχει ζητήσει το λόγο. Ε, ευχαριστούμε πολύ κυρία Μάρκας. Χάρηκα πάρα πολύ που ήρθατε να μας μιλήσετε. Ε, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη πιστεύω ότι θα μπορέσετε να προωθήσετε την πολιτική συνοχή στην Ιταλία. Συχνά έχουμε συζητήσει την κατεύθυνση της πολιτικής συνοχής. Τώρα μπορούμε να έχουμε ένα εξαιρετικό παράδειγμα και ίσως να φροντίσουμε στο μέλλον να ε, έχει πολύ μεγαλύτερη επικουρικότητα η πολιτική συνοχή. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση που κάνατε. Έχετε απόλυτο δίκιο για τη... τους λόγους που παρουσιάσατε σχετικά με την Ιταλία. Παρά τα αυτά, μια ερώτηση. Η Ιταλία δεν είναι μόνο η χώρα που έχει το χαμηλότερο ποσοστό χρήσης των ταμείων, αλλά έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό σφάλματος όσον αφορά τις δαπάνες αυτό δεν είχε άμεση σχέση με την συνδιαχείριση, αλλά με έναν ασαφή κανονισμό, δηλαδή την υποβολή προσφορών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Σε σχέση με αυτό που θα δούμε με την αιρεσιμότητα, εκ των προτέρων αιρεσιμότητα στο τέλος, στο μέλλον. Υπάρχει δυνατότητα όταν θα έχει ανατεθεί ένα έργο να είναι ξεκάθαροι κανόνες ή θα συνεχίσει να υφίσταται αυτή η δαμόκλειος αυτη η δαμοκλειο σπαθη με τα σφάλματα που θα συνεχίσουν να γίνονται σε βάρος των περιφερειών. Θα ήθελα να μου απαντήσετε. Να συγκεντρώσουμε δύο-τρεις ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ο κ. Γκουτμάνης. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. έχω να ρωτήσω ε, κάτι σε σχέση με τα έκτακτα μέτρα που πιστεύω ότι πρέπει να προωθήσετε. Βλέπουμε ότι το ποσοστό απορρόφησης της Ιταλίας το Ταμείο Συνοχής μέχρι φέτος 1η Δεκεμβρίου είναι δύο φορές χειρότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 18% και το πρόβλημα είναι ότι αυτή η κατάσταση σε όλη τη διάρκεια του 2011 έχει παγώσει. Μια πολύ μικρή αύξηση, 1,5% ε, μεταξύ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Όταν βλέπουμε το κοινωνικό ταμείο, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, αλλά και πάλι είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο. Και η ερώτησή μου είναι, δεν έχετε τόσο μεγάλο έλλειμμα το 2011 και το 2012. Εξακολουθεί η κυβέρνηση να προσπαθεί να ε, διατηρήσει χαμηλό το έλλειμμα μη προσφέροντας συγχρηματοδότηση ή το πρόβλημα βρίσκεται συνολικά στα έργα. Δηλαδή ότι οι δικαιούχοι δεν μπορούσαν να υποβάλουν οι υγιή έργα, προτάσεις που να μπορούν να πραγματοποιηθούν και άρα δεν είχε άλλη λύση παρά να μην συγχρηματοδοτήσει η κυβέρνηση. Αν δούμε και το, την περίοδο 2000-2006, την προηγούμενη δημοσιονομική προοπτική, η Ιταλία μέχρι το μέσο του, της χρονιάς φέτος δεν έχει μπορέσει να καλύψει το ένα δις ευρώ που είναι το 2006 συν 5. Ευχαριστώ, Elizabeth Σρέτερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Μπάρκα, χαίρομαι πολύ που έχετε τώρα τη δυνατότητα να θέσετε, στη, δοκιμάστε στην πράξη τις θεωρίες σας. Θα δούμε αν υπό τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει η Ιταλία θα μπορέσει να αποδειχθεί η θεωρία την ισχύ τη. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι οι καινοτομίε στα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τι ε, ε, μειονεκτικέ περιοχές, μια σειρά από έργα είχαν πρόβλημα και διερωτήθηκε κανεί αν, μπορούσαν, να είχαν βιωσιμότητα. Και τώρα εσείς προσπαθείτε να αλλάξετε τελείως ε, κατεύθυνση υπό δύσκολες συνθήκες και σας έχετε τον απόλυτο σεβασμό μου. Παρακολουθούμε πολύ στενά τις προσπάθειές σας να δούμε αν θα επιτύχουν. Διότι συνολικά πάντοτε παρακολουθούσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον τις θεωρίες σας και όλοι θέλουμε να δούμε μία περιφέρεια επιτέλους όπου να ισχύσει αυτό το result-oriented implementation στην πράξη. Η διαδικασία φυσικά θα είναι δύσκολη. Εσείς καταφέρατε να λάβετε υπόψη σας το άλλο σκέλος της θεωρίας σας. Θυμάμαι ότι είχατε πει ότι αυτό είναι σημαντικό και θέλεις, έχετε εμπλέξει τις περιφέρειες σε αυτή την προσπάθεια που κάνετε για τη μεγάλη στροφή οι τοπικές αρχές. Υπάρχει η αρχή της εταιρικής σχέσης, αλλά εξ όσων γνωρίζω με, από τις επαφές με τους Ιταλούς εταίρους, ελάχιστα έχουν εμπλακεί οι κοινωνικοί εταίροι, οι εταίροι στον τομέα του περιβάλλοντος, στο τομέα της ε, ε, εμπλοκής των φύλων, πρέπει να συμμετέχουν σε ε, ομάδες εργασίας, στην Επιτροπή Παρακολούθησης, να... αυτό είναι αυτό που προβλέπει ο κανονισμός. Θα το υλοποιήσετε και αυτό, θα το εφαρμόσετε. Θεωρώ ότι αυτό είναι το άλλο σκέλος της θεωρίας σας που είναι σημαντικό, πρέπει να εφαρμοστεί και αυτό είναι πιο δύσκολο να, να εμπλακούν οι οργανώσεις βάσει σε αυτές τι δύσκολες συνθήκες, αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι σκοπεύετε να κάνετε, τι πρόκειται να κάνετε. Υπουργό Πάρκα. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε. Ναι, έτσι είναι. Πάρα πολύ σημαντικό ο ρυθμός ή τέλο πάντων το ποστό των σφαλμάτων. Είναι κλασικά θέματα αυτά. Και έτσι αυτό είναι ένα καμπανάκι που χτυπάει, προειδοποίηση. Και έχουμε αυτή την κακή παράδοση να τα κάνουμε όλα τελευταία στιγμή. Όλα αυτά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν και έχετε δίκιο στο βιβλίο, το καταλαβαίνω. Η αιρεσιμότητα είναι πάρα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό για, για το ακριβώς όπως ορίζεται και ως πάρτιμα 4 θα πρέπει να δούμε. το πώς θα ληφθεί υπόψη και συνειδητοποίησε επιστρέφοντας στη χώρα μου ότι οι δημόσιες συμβάσεις και οι διαγωνισμοί δεν είναι βέβαια το μόνο σημείο που πάσχει από τόσα ασφάλματα, αλλά έχετε δίκιο στον την ρεσιμότητα. Και θίξατε το γιατί βρίσκεται τόσο πίσω η Ιταλία. Και τα δε στοιχεία που έχουμε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού και έχω εδώ κάποια στοιχεία, θα σα τα αφήσω, είναι στα ιταλικά, το άλλο και θα σα αφήσω είναι στα αγγλικά, το το Κοινοβούλιο και μετά από μία τριετία. Τι λέει, α, 2010. Ε, μετά από μία τετραετή περίοδο προγραμματισμού είμαστε στο 7,4%. Τώρα είμαστε στο 12% και ήταν 14,4% η υπόλοιπη Ευρώπη. Επομένως διατηρήθηκε αυτή η διαφορά του διπλάσιο, αλλά ε, έχει σημασία το ότι οι ίδιες χώρες ήταν στο ίδιο ποσοστό. Πριν από 7 χρόνια ήμασταν στο 16 και 16,6 και η υπόλοιπη Ευρώπη, πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Οι χώρε που ήταν τώρα 14,4 ήταν στο 21,3. Αυτό τι σημαίνει, ότι όλοι μας επιδεινώσαμε τις επιδόσεις μας. Εμείς όμως πολύ περισσότερο από τους άλλους. Τι είναι αυτό το θέμα σηματοδότηση και θέμα ποιότητα των προγραμμάτων. Η ποιότητα είναι πρόβλημα. Γιατί το θέμα είναι πού πάνε τα χρήματα που δαπανώνται. Τι μαθαίνουν οι ψηφοφόροι, τι μαθαίνει ο κόσμος, τοπονύμια και το πόσα χρήματα δαπανώνται. Όμως όλες αυτές τις ανακοινώσεις δεν κινητοποιείται κανείς γιατί δεν υπάρχει πίεση στη δίκηση για να κάνει κάτι. Όμως έχουμε αυτό το εσωτερικό σύμφωνο σταθερότητος. Και η συγχρηματοδότηση έχει άμεση σχέση με τις δαπάνες που γίνονται. Γι' αυτό και λέμε για αυτό το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που θα πρέπει να αντισταθμιστεί στα πλαίσια του προγράμματος σταθερότητας όπως μας είπε και η Κομισιόν. Τελευταίο τώρα. Α, μάλιστα. Αυτά που σας είπα πέρασαν από λεπτομερείς διαβουλεύσεις με τις περιφέρειες της χώρας και τους ευρώμους. Είχαμε την κλασική αντίληψη της πρωτεύουσα. η Ρώμη ήθελε φυσικά τις βασικούς άξονες, όμως οι περιφερειακές διοικήσεις ε, είχαν διαφορετική ιδέα, διαφορετική άποψη. Και για, για αυτούς ε, που κάθε μέρα πάνε στην τη δουλειά τους και ξαναγυρίσουν. Και είχαμε συμμετοχή με το facebook, με το twitter, όλους οι οποίοι βγήκαν σε εφημερίδες και είπαν ναι λέτε για τους βασικούς άξονες, τι θα γίνει όμως με τα άλλα δρομολόγια τα μικρότερα. και σε κάποιο κρατικό κτίριο στην Ρώμη. Συνεδριάσαμε, βρεθήκαμε με των περιφερειών και τα συζητήσαμε. Και έτσι δώσαμε σάρκα και οστά σε αυτές τις ιδέες. Τώρα η συνεργασία, η εταιρική σχέση. Τα πράγματα κάπως είχαν παγώσει, εμείς τα ξεπαγώσαμε. Οπότε ξαντήθηκαμε με τους εμπλεκόμενους Βέβαια είχαμε εκείνη τη μέρα απεργία των συνδικάτων. Με έναν κληθεί γενική γραμματής τους και τελικά υπήρξε ευρεία στήριξη και εγκρίθηκαν αυτά τα οποία προτείναμε από το Κοινοβούλιο. Και επίσης ανεβίωσαν κάποια μέτρα για τους ηλικιωμένους. και αυτά τα κάνουμε με μια αυθεντική μέθοδο συνεργασίας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω και εγώ κύριε Υπουργέ. Σας απευθύνομαι στην κοινή μας ε, μητρική γλώσσα, διότι και η γλωσσική αναγνώριση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας μεγάλης μάχης που δίνουμε ε, εδώ έτσι ώστε να μην πρέπει να απαρνηθούμε και αυτό το δικαίωμα κάποια στιγμή του να μπορούμε να εκφραζόμαστε στη μητρική μας γλώσσα. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε μιλήσατε για το σχέδιο το οποίο συμφωνήθηκε πρόσφατα με ορισμένες Ιταλικές περιφέρειες, ιδιαίτερα στο Νότο στη μεσημβρινή Ιταλία και από όσο γνωρίζουμε δεν θα πρέπει η περιοχή του Μέτζο Τζόρνο να χάσει σημαντικούς σπόρους. Και διατρέχουμε αυτό το κίνδυνο όπως πολύ καλά γνωρίζουμε. Καθότι δεν τηρήθηκε ο περιφερειακός προγραμματισμός. Νομίζω λοιπόν ότι δεν τηρήθηκε αυτός ο περιφερειακός προγραμματισμός διότι παράλληλα με την χρηματοπιστωτική κρίση είχαμε χαμηλότερη εισρωή πόρων προς περιφέρειες ε, μέσα στα πλαίσια του συμπληρωματικού χαρακτήρα των ε, μέτρων αυτών και η παρέμβασή σας αφορά την επαναδιαπραγμάτευση του εθνικού δίκτυ που μειώνεται από 50% σε 25%. Έτσι τουλάχιστον εγώ διαβάζω τα δεδομένα. Αν μπορείτε να με διορθώσετε, καλώς. Διότι από ό,τι φαίνεται έγινε επαναδιαπραγμάτευση της ε, συγχρηματοδότησης και γι' αυτό σας αποτείνω και αυτό το ερώτημα το οποίο απορρέει από στοιχεία τα οποία είδα και έζησα η ίδια γιατί έγινε λόγος για μείωση της συγχρηματοδότησης και βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την αλλαγή του κανονισμού, όπως έγινε για άλλες χώρες. Και βλέπουμε ότι ισχύει ήδη για άλλες χώρες. Αυτό λοιπόν είναι ένα ερώτημα προς εσάς. Μετά υπάρχει το θέμα το οποίο έχουμε δει πολλές φορές ως η Ιταλική αντιπροσωπεία. Δηλαδή είδαμε τους όρους που συνοδεύουν την μελλοντική, το μελλοντικό προγραμματισμό. Αυτή η πρόβλεψη αφορά έναν μεγαλύτερο έλεγχο, μια σοβαρή εποπτεία και θέλουμε να αποφύγουμε τα σφάλματα του παρελθόντος, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Υπάρχουν δυσκολίες εκπλήρωσης των στόχων, άρα πολύ σωστό το να υπάρχουν σοβαρότερες κυρώσεις και μεγαλύτερη αιρεσιμότητα όμως. Η μακροαιρεσιμότητα που συνοδεύει την πολιτική συνοχής με βάση τις παραμέτρους του Μάστριχτ και του Συμφώνου Σταθερότητας είναι μια ιδέα, αποτελούν μια ιδέα την οποία δεν συμμεριζόμαστε γιατί μας ενδιαφέρει πέρα από το γράμμα και το πνεύμα της πολιτικής συνοχής. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό δεν συνάδει με την πολιτική συνοχής και αλληλεγγύης που θα πρέπει να ισχύει. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω σε σχέση με μια πολιτική αντισταθμίσεων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να τηρήσουμε τους κανόνες και ως προς την εταιρική σύμβαση, νομίζω ότι ενισχύεται από την επιτροπή της, από την πρόταση της Κομισιόν. Γι' αυτό θα πρέπει να διατρανώσουμε τη θέλησή μας και έτσι να δώσουμε στις περιφέρειες μια μεγαλύτερη αυτονομία γιατί συμμερίζομαι την ανησυχία και της κυρίας Σρέτερ. Πιστεύω ότι αυτό το ενδεικτικό σχέδιο που μας προτείνεται κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, αφήνουμε το όλο θέμα στην κεντρική κυβέρνηση. Θα ήθελα να μου απαντήσετε επί των θεμάτων αυτών. Ευχαριστούμε. πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν επτά ομιλητές ακόμα, γι' αυτό θα ήθελα να επιταχύνετε τους ρυθμούς. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για τους ταλούς συναδέλφους, γιατί έχουμε τον Φαμπρίτσιο Μπάρκα εδώ. Ε, ο κύριος Σούτζας ζήτησε το λόγο. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω σας καλωσορίζω με, τη, με βάση τη νέα σας ιδιότητα και την πείρα σας. Ευπρόσδεκτες και οι ιδέες και οι προτάσεις σας. Είχαμε ζήσει ένα μεγάλο κενό μέχρι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια. Και εδώ και ένα χρόνο η Ιταλική κυβέρνηση δεν όριζε έναν, δεν διόριζε υπουργό για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Άρα δεν μας εκπλήσει το γεγονός ότι σήμερα δεχόμαστε αλλεπάλληλα χτυπήματα σε σχέση με τις ε, κεντρικές και περιφερειακές επιλογές. Είδα ότι προσδίδεται μεγάλη σημασία έτσι ώστε να μην χαθούν πόροι από τον τρέχοντα προγραμματισμό. Όπως όμως γνωρίζετε θα πρέπει να σκεφτούμε και το μέλλον, διότι έχουν ανοίξει όλοι τα χαρτιά τους και για τον προγραμματισμό της περίοδου 14-20. Μιλήσατε για μια ενισχυμένη συνεργασία με την Ένωση. Σας υποβάλλω λοιπόν μια ερώτηση. Μπορούμε να προωθήσουμε ενισχυμένη συνεργασία με το Κοινοβούλιο και να ορίσουμε το τετραγωνίδιο αναχώρησης. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα στοιχεία είναι αυτά που είναι. Μπορούμε όμως να συντονίσουμε τις προσπάθειες έτσι ώστε να ορίσουμε και μέτρα για το μέλλον, για ένα πλαίσιο έτσι ώστε όλες οι περιφέρειες και η Ιταλία να έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πόρους που είναι και η μοναδική που διαθέτουμε. Μετά έχουμε τη δυνατότητα εμβάθυνσης ε, αλλού. Αλλά αυτό σας το θέτω ως ε, πρωταρχική ερώτηση. Επίσης, μιλήσατε για τον κυβερνητικό προγραμματισμό, για τον επαναπροσδιορισμό και επανακατανομή των πόρων για τη μεσημβρινή Ιταλία, για το Μετζοτζόρνο. Η ερώτηση λοιπόν έχει ως εξής. Δεν υπάρχει πρόθεση να αντικαταστήσουμε αυτούς τους πόρους με κάποιους άλλους, δηλαδή να υπάρχει μία πολιτική πίστοση. Πρόκειται για ένα ηθικό ε, μέλημα της κυβέρνησης, έτσι ώστε να μην γίνει υποκατάσταση, γιατί τότε ε, θα χάναμε. Έχετε ορισμένες σχετικές ιδέες έτσι ώστε να προβάλλουμε ε, νέους πόρους οι οποίοι να υποκαταστήσουν τους υπάρχοντες. Θα ήθελα, λέει ο κύριος ε, Καρόνα, να σας συγχαρώ. Σας εκφράζω τις ευχές μου για τις νέες σας αρμοδιότητες. Κάτι που μας απασχολεί τα τελευταία χρόνια είναι να λάβουμε υπόψη ότι έχουμε χάσει εμπολή στην αξιοπιστία μας. Θα ήθελα να σας υποβάλω ορισμένες ερωτήσεις λοιπόν. Λυπάμαι που η Κωνσταντσε έφυγε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η θέση σας για την εισαγωγή της νέας ενδιάμεσης κατηγορίας. Η δεύτερη σκέψη έχει ως εξής. Όσον αφορά το ρόλο των περιφερειών. Ποια είναι η θέση σας ως προς το ε, εταιρικό, την εταιρική σύμβαση. Ε, διότι ζητάμε να εισαχθεί ως βασικό στοιχείο αυτή η σύμβαση, η εταιρική σύμβαση και ποιος θα είναι ο ευρωπαϊκός κώδικας που θα μας ε, διέπει. Αυτές είναι οι σκέψεις και οι ερωτήσεις μου. Θα απαντήσω και εγώ στην ερώτηση της κυρίας Ματσόνη στα Ιταλικά. Η επαναδιαπραγμάτευση της ε, συγχρηματοδότησης ανήκε σε μια διαφορετική κατηγορία από αυτήν ε, που ίσχυε μέχρι τώρα. Άρα θα μειώσουμε τον ε, δίκτυ συγχρηματοδότησης και μιλούσαμε για μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου ο δίκτυ συγχρηματοδότησης ήταν ο στόχος η χώρα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτούς τους πόρους για αποταμίευση ή για άλλους λόγους. Εμείς κάναμε άλλη επιλογή. Η Στάμπα έγραψε ότι η Ιταλία θα μειώσει τον δίκτυο από 50 σε 25. Την, ε, ως προς την κοινοτική χρηματοδότηση. Εμείς δεν το είπαμε αυτό. Εμείς ξεκινήσαμε από προγράμματα έχοντας ορίσει συγκεκριμένα προγράμματα για τους σιδηροδρόμους που χρειάζονται 10 χρόνια για να πραγματοποιηθούν, ποσοστοποιήσαμε τον δίκτυ συγχρηματοδότησης αφού αποφασίσαμε για τα προγράμματα. Άρα η μείωση δεν είναι η ίδια σαν να είχαμε περάσει από 50 σε 75, δηλαδή 8 δις. Δηλαδή ούτε καν ποσοστοποιήσαμε. Νομίζω ότι μιλάμε από, για 50, 54, 55. Μιλήσαμε για 1 δις 500 εκατομμύρια μέσα στα πλαίσια συγκεκριμένων προγραμμάτων. Εκτός από τα κοινοτικά ταμεία. Υπάρχει ένα ταμείο που αφορά τους σιδηροδρόμους, όπου ορίζει τα ποσά εκκίνησης για τους σιδηροδρόμους. Δεν μειώνεται το ποσοστό για τους κανονισμούς. Υπάρχει κίνδυνος ε, συγκέντρωσης. Όχι, γιατί όπως απάντησα και στη συνάδελφο της Γερμανίας, το θέμα συμφωνήθηκε με τις περιφέρειες και συζητήθηκε. Και μόνο οι σιδηρόδρομοι θα ανατεθούν στις κεντρικές αρχές. Διαφορετικά έχουμε περιφερειακά προγράμματα. Η κυβέρνηση διαδραματίζει το ρόλο που της αρμόζει. Δηλαδή εποπτεύει και συνοδεύει. Δηλαδή, εάν γίνονται παρεμβάσεις ε, για τα σχολεία, σε επίπεδο σχολείων, η κεντρική κυβέρνηση θα πρέπει να συντονίσει την κατάσταση. Αυτό αφορά και την ψηφιακή ατζέντα που εντάσσεται στην Ευρώπη 2020. Δεν ε, υφίσταται κανένας κίνδυνος. Λοιπόν, ως προς την ε, μακροαιρεσιμότητα γνωρίζετε τη θέση μας, γνωρίζετε μάλλον όχι τη δική μας, τη θέση της Ιταλίας. δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο τη συνοχή. Η Ιταλία παραβίασε την προσθετικότητα διότι περιέκοψε πόρους που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί. Τη στιγμή λοιπόν που τα λογιστικά μας στοιχεία δεν είναι σωστά, θέτουμε σε κίνδυνο την ίδια τη συνοχή. Άρα θα πρέπει να υπάρξουν και κυρώσεις για τις χώρες που δεν τηρούν τους όρους. Οι όροι όμως θα πρέπει να είναι οι κατάλληλοι όροι και θα πρέπει να είναι αναλογικοί. Δεν θεωρούμε λοιπόν ότι υπάρχουσα πρόταση είναι σωστή, διότι δεν τηρεί την αρχή της αναλογικότητας. Θα πρέπει λοιπόν να ορίσουμε άλλες αρχές. Θα επανέλθω στα αγγλικά. Όσον αφορά την περίοδο 2014-2020, θεωρώ ότι η Ιταλία πιστεύει στον θεμελιώδη σημαντικό ρόλο του κοινοβουλίου σας και γι' αυτό και χαίρομαι που το συζητούμε τώρα εδώ το θέμα και όσον αφορά τον ρόλο των περιφερειών νομίζω ότι αυτό το ταυτόχρονο της έγκρισης του λειτουργικού προγράμματος και των ε, συμβάσεων εταιρικής σχέσης τους δίνει των περιφερειών πάρα πολύ ε, σημαντικό ρόλο. Δεν υπάρχει εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Ταυτόχρονα γίνεται η απόφαση. Οπότε γι' αυτό και θέλουμε να υπάρχει ανοιχτή συζήτηση με την Επιτροπή και όχι ε, ξαφνικά να αποφασιστεί οτιδήποτε τεχνοκρατικά. Τώρα, όσον αφορά τις ενδιάμεσες περιφέρειες, όχι, δεν θεωρεί η Ιταλία ότι αυτό είναι σωστή μέθοδος, η βαθμιαία κατάργηση δεν είναι η καλύτερη λύση. Θέλουμε να συζητηθεί αυτό και με τα άλλα κράτη-μέλη. Κύριε Ντιάντζελης. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο και σας συγχαίρω για το νέο σας χαρτοφυλάκιο. Υπάρχει σωρία ερωτήσεων, αλλά εγώ θα περιοριστώ σε μία που θεωρώ ύψης της σημασίας. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, η ποιότητα των δαπανών γιατί μιλάμε για ποσά και αριθμούς, αλλά δεν μιλάμε για την ποιότητα της δαπάνης, διότι η καλή χρήση αυτών των δαπανών ορίζει και την ανάπτυξη και την εργασία μας, τις εργασιακές μας προσπάθειες, ποια μέσα προβλέπετε για να φτάσετε σε αυτό το στόχο που θεωρώ ε, στόχο κατά προτεραιότητα, δηλαδή η εύρυθμη ε, χρήση των ταπανών. Όλμπρεχτ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Πάρα πολύ χαιρόμαστε που είστε εδώ και με την νέα σας ιδιότητα, όμως βέβαια περισσότερο από τα τέλεια προβλήματα. Πέστε μας από την σημερινή σας θέση και βάση της εμπειρίας σας, τι βλέπετε για το μέλλον. Έχω πάρα πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει να σας υποβάλω. Στο εγγραφό σας υπάρχει κάτι το οποίο παρακαλώ εξηγήστε μου. Τι είναι τα εθνικά κέντρα που έχουν την αρμοδιότητα. Θυμάμαι. Στην πρωταξιακή περίοδο τα λέγαμε στις διαφορετικές ε, επιτροπές. Τότε είχατε την ελεγκτική αρμοδιότητα και τώρα θέλετε η Επιτροπή να διαμορφώνει τις προτάσεις. Αυτό θα ισχύσει και για το μέλλον ή απλώς αυτό είναι προσωρινό λόγω κρίσης. Άλλη ερώτηση. Τι λέτε ως Υπουργό για το κοινωνικό πλαίσιο στήριξης. Τι είναι, είναι αυτές οι κατεχώρες αρμοδιότητες και πράξεις. Τι λέτε, τι πιστεύετε. Τώρα και κάτι άλλο. Η θεματική συγκέντρωση. Τι συνέπειες έχει για σας ως Υπουργό σήμερα. Θεωρείτε ότι αυτό είναι θετικό. Θα πρέπει να έχει περισσότερη ευελιξία, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να αποφασίσουν. Αν θέλει τώρα το λόγο και ο κύριος Λάμπερτ, οπότε βάζω εδώ τελεία. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Και εγώ χαίρομαι για την παρουσία του κυρίου Μπάρκα, τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια και θυμάμαι όταν ε, είχαμε την διακυβέρνηση υπό τον πρώτη μας είχατε εκπροσωπήσει για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές μέχρι το 2013. Μιλάμε λοιπόν για ένα νέο ρόλο των Ιταλικών αρχών και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε δύο βασικά θέματα. Το πρώτο αφορά την έλλειψη τα τελευταία χρόνια ενός ε, πλαισίου, εθνικού πλαισίου στήριξης έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές και να ορίσουμε και τις, την αυτονόμηση των ε, περιφερειών. Νομίζω ότι η εταιρική σύμβαση μπορεί να αντικαταστήσει το εθνικό σχέδιο για το 2000 μέχρι το 2015. Αυτό θα το ανακτήσουμε στρατηγικά έτσι ώστε να έχουμε μία περιφερειακή διακυβέρνηση. Το δεύτερο θέμα αφορά το στρατηγικό πλαίσιο. για να υπάρχουν διαπεριφερειακές συμφωνίες. Γιατί πολλές φορές μιλάμε για προγράμματα όπου θα πρέπει να υπάρχει μία συνδεσιμότητα μεταξύ τους. Δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω. Ενώπιον της κρίσης χρησιμοποιήσαμε το ΕΚΤ για τις περιφέρειες έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε μικρές επιχειρήσεις με την επιδότηση του ΕΚΤ. Όμως η αιρεσιμότητα που σήμερα θα αποτελέσει σημαντικό στοιχείο ίσως ε, προβάλλει νέες, ε, νέους κοινωνικούς θύλακες έτσι ώστε να καλύψουμε ορισμένα κενά. Άρα η αιρεσιμότητα σε σχέση με χώρες όπως η Ιταλία ή άλλες όπου υπάρχει έντονος τοπικός χαρακτήρας θα δοθούν χρήματα για τις διαρθρωτικές προσαρμογές σε περιφερειακό επίπεδο. Δηλαδή στο νέο προγραμματισμό θα υπάρχει ερεσιμότητα σε σχέση με το εθνικό αρνητικό outlook ή σε σχέση με το θετικό περιφερειακό outlook. Θα πρέπει να δούμε δηλαδή κατά πόσο υπάρχει η αρχή της αναλογικότητας και της επικουρικότητας που θα ισχύει. Επίσης θα πρέπει να ορίσουμε καλύτερα και να κατανοήσουμε ποιες είναι αυτές οι διαδικασίες που θεωρητικά είναι πολύ καλές αλλά είναι άχρηστες στην πράξη διότι ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε τις ε, διαδικασίες για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα όλα τα ταμεία και ιδιαίτερα το ΕΚΤ. Η κυρία Τόιρερ. Ο κύριος Τόιρερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπάρκα που ήρθατε. Ως ε, εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο ψήφισε την έκθεσή μου για τα ποσοστά απορρόφησης και τα προβλήματα της απορρόφησης. Μελετήσαμε τα προβλήματα και τα αίτια της χαμηλής απορρόφησης σε κάποιες περιφέρειες και μελετήσαμε τις βέλτιστες πρακτικές κάποιων. Είναι σκάνδαλο που δεν μπορούν κάποιες περιφέρειες να απορροφήσουν τα κονδύλια. Δεν είναι μόνο θέμα στη χρηματοδότηση, είναι και θέμα δημιουργίας δυνατοτήτων, είναι θέμα της λειτουργίας και της ε, ισχυρής τοπικής και περιφερειακής κυβέρνησης και γι' αυτό ζητήσαμε, για, ζητήσαμε αποκέντρωση και κατάρτιση. Επειδή πασίγνωστος εδώ στις Βρυξέλλες αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την έκθεση Μπάρκα που έχετε υποφάλει. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, λόγω της εμπειρίας που φέρετε από την Ιταλία, τα διαρθρωτικά ταμεία και το, το Ταμείο και, και το Ταμείο Συνοχής θα μπορούσε να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη σταθεροποίηση της κατάστασης όπως είναι τώρα, όχι μόνο στο πρόβλημα του κρατικού χρέους και των εντάσεων της Ευρωζώνης. Πιστεύω ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να, ε, τις προσπάθειες των Ταμείων Συνοχής και Διαρθρωτικών Ταμείων στα θέματα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, κυρίως σε κάποιες περιφέρειες. Ποια είναι η άποψή σας σε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Ευχαριστώ τον τελευταίο λόγο θα τον έχει ο Λάμπερτ Φανίστεροι. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Μπάρκα, χαιρόμαστε που μας ακούτε και πάλι από αυτή τη θέση. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, στην έκθεση Μπάρκα αναφερθήκατε ε, στις συμβάσεις που θα πρέπει να γίνονται. Η δική σας τώρα προσέγγιση είναι καλό παράδειγμα αυτού το οποίο εννοούσατε στην έκθεσή σας. Γιατί χρειάστηκε να αναδιοργανώσετε και να αλλάξετε κάποια πράγματα. Είναι αυτού του είδους οι συμβάσεις αυτές οι οποίες προτείνετε στην έκθεσή σας. Και δεύτερο ερώτημα. Αν δω τις προτεραιότητές σας, κάτι μου λείπει. Κάτι μου λείπει. Το κομμάτι που αφορά την ενέργεια. Αν μιλάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2020, ήδη εκεί είμαστε θεώρηση προτεραιοτήτων. Μια μεγάλη ευκαιρία για την ε, Νότια Ιταλία και δεν το βλέπω αυτό. Για ποιο λόγο. Τρίτη ερώτηση. Σε σχέση με αυτά που συζητάμε. Πολλά χρήματα μπορούν να δαπανηθούν στην παιδεία. Είπετε ότι το θέλετε, θέλετε να γίνει αυτό προτεραιότητα. Αν δεν αλλάξει η αγορά εργασίας, αν δεν υπάρξει ευελιξία, μπορούμε να δαπανίσουμε χρήματα και να πιστεύουμε ότι θα αποδώσουν. Αλλά υπάρχει κάτι παραπάνω. Η κυβέρνησή σας έχει διαφορετική προσέγγιση. Αν δούμε την, ε, εκ των προτέρων τα αποτελέσματα, πιθανά, εκ των προτέρων τα πιθανά αποτελέσματα Πώς το βλέπετε, είναι η συνολική προσέγγιση της κυβέρνησής σας αυτή. Μπορείτε να μας μιλήσετε από αυτό. Ευχαριστώ. Φαμπρίτσιο, έχει το λόγο. θα, θα συγκεντρώσω όλες τις ερωτήσεις που αφορούν την Ιταλία καταρχήν και μετά θα αναφερθώ στο μέλλον. Το πώς περιμένουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα. Η ποιότητα είναι ζωτική σημασία ζήτημα και σκοπεύουμε να το καταλάβουμε προκαταλαμβάνοντας ε, την χρήση κάποιων μέσων του νέου κανονισμού. Έχουμε ένα σχέδιο δράσης που θα προτρέξει κατά κάποιο τρόπο. Απαντώ εν μέρη στη δική σας ερώτηση. Είναι μια σύμβαση η οποία γίνεται με όλους περισμούς που γίνεται, την ώρα που γίνεται υπάρχει και η λειτουργία. Προκαταλαμβάνουμε λοιπόν κάποια νέα στοιχεία, προτρέχουμε και αυτό εν, μέρη είναι οι δείκτες αποτελέσματος που θα συμπεριληφθούν στο σχεδιασμό αλλά και στην αποτελεσματικότητα. Δηλαδή θα βάλουμε ε, χρήματα για τα σχολεία και θα, θα δούμε αυξάνουν οι μαθηματικές δεξιότητες των μαθητών στην πράξη ή απλώς πληρώνουμε καλύτερα τους δασκάλους. Το θέμα της προτεραιότητας και έρχομαι στην τελευταία ερώτηση γιατί είπα ότι θα κεντρώσω τα θέματα της Ιταλίας. Η ενέργεια δεν υπάρχει γιατί ήδη υπήρχε, υπήρχε πρόγραμμα ενέργειας που στην Νότια Ιταλία είχε δώσει αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Μιλάμε για τα άσχημα αλλά υπάρχει και αυτό. Αν δεν, αν δεν κάνω λάθος η Ιταλία έχει αυτή τη στιγμή ένα ποσοστό ε, ε, χρήσης ε, ίδιας ενέργειας που δεν προέρχεται από ανανεώσιμες και από υδροελεκτρικές πηγές διπλάσιο από ό,τι στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Και το τελευταίο για την αγορά εργασίας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μάλλον το πακέτο για τα σχολεία. Ένα κομμάτι του αφορά την ποιότητα των σχολείων. Δεν θα έπρεπε να γίνεται τέτοιο θέμα ε, ε, σε μια χώρα που είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρά τα αυτά, κάποια, η ποιότητα κάποιων σχολείων στην Νότια Ιταλία απέχει παρασάγκας από το επιθυμητό και δεν μπορεί κανείς να ζητήσει από αυτά τα, σχολεία, από αυτά τα παιδιά να μην μπουν στο οργανωμένο έγκλημα, να, κάνουν, να σέβονται τους νόμους κλπ. Έχουμε 40 100 των παιδιών του Νότου που είναι κάτω των, του επίπεδου της πίζα στα μαθηματικά. Και είναι εκτός δηλαδή. Δηλαδή δεν θα μπορέσουν ποτέ να συνομιλήσουν με τους συμμαθητές τους στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά υπάρχει και ένα κομμάτι που αφορά αυτό που θέσατε κι εσείς, είναι η μετάβαση από το σχολείο στην αγορά εργασίας. Κάποιες νέες πρωτοβουλίες εφαρμόζονται με το σχέδιο αυτό που ελπίζουμε ότι τελικά θα χρησιμοποιηθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Σκοπός του Υπουργού Παιδείας και Έρευνας είναι κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες να χρησιμοποιηθούν ως πρότυπα για την ε, κανονική πολιτική. Αυτό που σας έλεγα πριν, μαθαίνουμε μέσω μιας εδαφικής πολιτικής σε, με πιθανότητα να, την, να καλύψουμε και, το, και τη Βόρεια Ιταλία. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον, τι εννοούμε όταν λέμε εθνικά κέντρα ε, National Competence Centers, είναι μια γενική διεύθυνση της κεντρικής διοίκησης. Ας πούμε, ε, ε, στο, στο, στο πεδίο της παιδείας. Υπάρχει ε, μια γενική διεύθυνση ας πούμε πολύ καλή παιδείας και χαίρει μεγάλου σεβασμού γιατί είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να είναι ένας φορέας, ένας οργανισμός. Ο οργανισμός συγκοινωνιών είναι εξαιρετικός, πάει πολύ καλά, έχει πολλούς μηχανικούς και θα θέλαμε να ασχολούνται περισσότερα ε, με τον Νότο γιατί έχουν επικεντρωθεί στο Βορρά ε, στρέφουμε την προσοχή αυτών των ε, ισχυρών φορέων στην περιοχή που δεν τους έχει απασχολήσει μέχρι τώρα. Είναι δημόσια τα κέντρα αυτά, εντός των διοικήσεων, εντός των οργανισμών, ε, των δημοσίων οργανισμών κλπ. Τώρα, η επικουρικότητα. Θα πειραματιστούμε και ελπίζω να μπορέσετε να μας ελέγχετε. Εγώ το βλέπω ως εξής κατανομή ευθυνών στις στρατηγικές επιλογές που δεν θα σταματούν τη στιγμή της συγγραφής του, της σύμβασης. Βλέπω μια συνέχεια με αυτά που κάναμε με την Τανούτα όταν συζητούσαμε τα διάφορα θέματα. Όταν μιλάμε για, δύναμη, για ομάδα δράσης, μιλάμε για μόνιμη ομάδα δράσης όπου η Κομισιόν δεν θα διατηρεί την ευθύνη θα αφήσουν, θα επιτρέψουν να τους ε, αμφισβητήσουμε. Θα έχουμε λοιπόν και κάποιους εμπέρους από τις Βρυξέλλες, ε, μυρογνώμες από τις Βρυξέλλες που θα συνεργαστούμε με τη Σαμπίνα και την Ιταλική ομάδα. Μιλάμε για μια στρατηγική, όχι για διαχείριση. Και αυτοί θα διατυπώσουν την ε, έλλειψη ικανοποίησή τους για κάποιους δείκτες, αλλά όχι σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο αλλά θα προκαλέσουμε την Επιτροπή να μας δώσει κάτι το οποίο θα αποτελέσει πρόκληση για μας. Το είναι δύσκολο αυτό, γιατί έχετε ε, κάτι επιτάπητος και τους καλείτε να αντιδράσουν ταχύτερα. Έτσι είναι. Αυτό είναι δύσκολο. Ε, μπαίνουμε στο προσκήνιο για να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Ναι, πραγματικά είναι ένα είδος προτύπου. Το κοινό στρατηγικό πλαίσιο. Εξακολουθώ να ανησυχώ για το κίνδυνο. Γι' αυτό πρέπει να με η Ιταλία έχει μια ιδιαίτερη θέση μοναχή. Είμαστε μόνοι μας γιατί πιστεύουμε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να το συντάξει. Γιατί ε, αλλιώς εμείς θα καταλήξουμε σε κάποιο συμβιβασμό που θα δώσει ένα έγγραφο το οποίο δεν θα ε, είναι αποτελεσματικό. Εγώ στο τελευταίο συμβούλιο είπα, λέμουνα μόνος μου, ότι η Ιταλία πιστεύει ότι πρέπει να γίνει έγγραφο της Κομισιόν, να παραμείνει έγγραφο της Κομισιόν, να βρεθεί μια μορφή πρέπει να, ενισχυ... να υποστηριχθεί, να γίνει endorsed από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Είναι κάτι που μας πρότειναν να συνδυάζει την ε, νομιμότητα και την ε, ισχύ. Τώρα, όσον αφορά την θεματική συγκέντρωση, όπως έχουν αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην πρόταση, είναι πολύ άκαμπτο αυτό. Είναι πολύ επικίνδυνο ε, να πει κανεί ε, στην Καλαβρία που φτάνει που εσείς θέσατε. Ναι, στην Καλαβρία όμως δεν σημαίνει ότι θα στέλνουμε χρήματα σε όλα τα πανεπιστήμια, εκτός από δύο πανεπιστήμια στα οποία αξίζει να χρηματοδοτηθούν. Αν έχουμε υπερβολικά πολλούς πόρους και δεν απορροφώνται, πάνε χαμένοι. Στην Καλαβρία το θέμα της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας πρέπει να αντιμετωπιστεί με την επαναδημιουργία του κοινωνικού συμβολέου μεταξύ πολιτών και κράτους. Είμαστε 20 χρόνια πίσω. Αυτό είναι πρόβλημα, είναι παγίδα. Δεν μπορεί κανείς να κάνει άλματα. Σε κάποιες πόλεις μπορεί, αλλά δεν μπορεί κανείς να ζητήσει συνολικά από την Καλαβρία να κάνει τεράστιο άλμα και να ξοδέψει χρήματα σε τέτοια καινοτομία. Τι κάνει κανείς ε, τελικά. Θα κάνουν ε, προτάσεις σε επιχειρήσεις που είναι εκτός και δεν γνωρίζουν τίποτα, ούτε έρευνα ούτε τις επιχειρήσεις. Με ανησυχεί πάρα πολύ η πρόταση της Επιτροπής όπως έχει συνταχθεί. Βρίσκω την πρόταση του Κοινωνικού Ταμείου πιο λογική γιατί περιέχει μεγαλύτερη ευελιξία. Δεν ότι το έχουμε αποφασίσει, αλλά ο τρόπος σκέψης του κοινωνικού ταμείου όπου οι επιλογές θα γίνουν ε, θα υπάρξει συγκέντρωση, αλλά ε, η επιλογή για το επιτύνος θα επικεντρωθούμε, θα αφαιθεί στις περιφέρειες. Είναι πολύ ε, λογικό και καλό. Ζητώ συγγνώμη γιατί συνήθως μου αρέσει τόσο πολύ εδώ και ξεπερνώ το χρόνο μου. Στο, περιφερειακό, στο διαπεριφερειακό πρόγραμμα ναι, αλλά η δική μας εμπειρία δεν ήταν πολύ θετική, γιατί δεν ήταν απόλυτα σαφές ποιος ήταν επικεφαλής, ποιος ήταν υπεύθυνος. Είναι ένα ζήτημα εδώ με τα διαπεριφερειακά προγράμματα. Ναι, αλλά. Δηλαδή είναι η απάντησή μου, ναι, αλλά. Τώρα, η εισαγωγή της αιρεσιμότητας ε, θα μας κάνει να τα βλέπουμε εκ των προτέρων εξάντε και όχι εξπόστο τα πράγματα. Συμφωνώ, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε κάποια ευελιξία γιατί κανείς δεν ξέρει τι θα προκύψει. Και η Βόρεια Ιταλία αυτή τη φορά είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τους πόρους αυτούς ευέλικτα και αυτό ήταν πάρα πολύ μεγάλη τύχη για όλους μας. Αυτά. Ευχαριστώ. Um, ευχαριστούμε. Και με αυτό τα οποία μας είπατε ολοκληρώνουμε την ανταλλαγή απόψε με τον ε, Υπουργό, τον κύριο Φαμπρίτσιο Μπάρκα και εκ μέρου όλων θα πρέπει να σας πω ότι σας ευχαριστούμε και εκτιμούμε πάρα πολύ και τώρα τα όσα μας είπατε για το σχόλιο στην Ιταλία και για όσα θα κάνετε στο μέλλον γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με τον κανονισμό τον οποίο συζητούμε και από ό,τι γνωρίζουμε είναι διαιρημένο σε πολλά θέματα το Συμβούλιο. Και ευχαριστούμε που μας μιλήσατε τόσο λίγα σήμερα, πολύ σημαντικό για μας. Όποτε θέλετε κάτι να πείτε, μια που τώρα πειραματίζεστε και αν δείτε κάποια συμπεράσματα που είναι και για μας χρήσιμα να τα ακούμε. Όποτε θέλετε. Είστε ευπρόσδεκτος. Καλή επιτυχία, καλό κουράγιο για την κυβέρνηση του κυρίου Μόντι, για το έργο όλων των υπουργών, ελπίζουμε να τα καταφέρει η Ιταλία. Θα θέλαμε πάρα πολύ η πολιτική της συνοχής να σας βοηθήσει να βγείτε από τα διέξοδα. Καλά Χριστούγεννα.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 που το προγραμματίζουμε εδώ και δύο χρόνια είναι το ΕΠ και άλλα κριτήρια τη πολιτική για τη συνοχή. Και έχουμε τέσσερι εμπειρογνώμονε εδώ. Και η γραμματεία μα λέει να προχωρήσουμε όπω λέει η λογική. Ξεκινούμε με τον καθηγητή Γιάτσεκ Σάχτα που μας λέει για το πώς γίνεται η μέτρηση της ανάπτυξης σε σχέση με την πολιτική της συνοχή. Παρακαλώ να λάβουν υπόψη οι ομιλητέ ότι έχουμε μία ώρα και ένα τέταρτο. Αλλά θα πρέπει να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε χρόνο για συζήτηση, διευκρινήσει κλπ. Καθηγητά, έχετε το λόγο. Χωρί μικρόφωνο. Σα ευχαριστώ που με καλέσατε και θα προσπαθήσουμε να όσο γίνεται πιο σύντομος. Βλέπετε εδώ τα πιο σημαντικά αυτά τα σημεία τα βασικότερα σημεία του εθνικού λογαριασμού. Αυτά ξεκίνησαν από έναν μεγάλο διανοητή και τώρα τα επεξεργαζόμαστε και στην Ευρώπη και έχουμε εδώ πέρα τρεις διαστάσεις, την οικονομική, την κοινωνική και την εδαφική. Αυτά είναι η σύλληψη, η αντίληψη της συνοχής στην συνθήκη της Λισαβόνας. Ξεκινούμε από με την οικονομική πτυχή που είναι το ΑΕΠ και αυτό θεωρείται πάρα πολύ βασικό κριτήριο μέτρησης. Ε, κοινωνικό κριτήριο είναι το επίπεδο της, ε, του, το ποστού της ανεργίας αλλά και της απασχολησιμότητας και το εδαφικό κριτήριο ε, εδώ έχουμε προχωρήσει λιγότερο είναι η προσβασιμότητα, ο χρόνος της διαδρομής που πρέπει να γίνει. Αυτά. Και ναι και όχι όσον το ΕΠ. Βασικά θέματα. Ότι πάνω κάτω πρόκειται για ένα αντικειμενικό κριτήριο ε, εκτίμησης, αξιολόγησης της ε, παραγωγής, αλλά όχι της ευημερίας. Για κάποιο κράτος, για κάποια περιοχή. Αν πρέπει πάντως να συγκρίνουμε χώρες ή περιφέρειες, πρέπει να διαπιστώσουμε τι αναπτυξία έχουν, τότε είναι το καλύτερο κριτήριο. Και υπάρχουν πάρα πολλές απλουστεύσεις σχετικά με οικονομικές δραστηριότητες. Και θα μπορούσε ευκόλως να αποδειχθεί ότι είναι πάρα πολύ επιλεκτικό αυτό το κριτήριο αν είναι κάτι το οποίο αμείβεται, μετράει, αν όχι δεν μετράει. Επίσης είναι θέμα ε, βεληνικούς, είναι κάτι το οποίο ωφελεί ή όχι το περιβάλλον. Και πρόκειται επίσης και για την παραοικονομία στους εθνικούς λογαριασμούς. Επίσης είναι και το θέμα της ε, στρατιωτικής πολεμικής βιομηχανίας, αν μετράει. Επίσης ε, υπάρχουν προβλήματα συγκρισιμότητας μεταξύ των διαφορετικών ε, περιοχών, διαφορετικά επίπεδα τιμών. Και για να υπάρχει συγκρισιμότητα συνήθως ε, χρησιμοποιούμε την αγροστική δύναμη. Και σε δαφική κλίμακα προσπαθούμε να συγκρίνουμε και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο χώρας. Οπότε έχουμε τις περιοχές ΝΑΤΣ 2 και ΝΑΤΣ 3. Οπότε τα αποτελέσματα διαφέρουν πάρα πολύ. Σε σχέση με το έδαφος, την, περιοχή ή τον πληθυσμό. Προκύπτουν κάποιες ποιότητες αποτελέσματα. Να εδώ βλέπετε εδώ αυτόν τον χάρτη που είχαμε κατά νου σε σχέση με την τελευταία έκθεση για την συνοχή. Το ΕΠ κατά κεφαλή. Με κριτήριο την αγοραστική δύναμη. Αυτό το γράφημα προέρχεται από την, Αυτό ο χάρτης του πάντων από την Παγκόσμια Τράπεζα. Βλέπετε εδώ πέρα το ΕΠ ε, ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Βλέπετε τα Ιμαλάια είναι οι Βρυξέλλες. Μετά ακολουθεί αμβέρς αυτό. Είναι το αντίστοιχο για την Πολωνία. Μπορείτε να δείτε ότι τα πάει πάρα πολύ καλά η Βαρσοβία και στις άλλες αστικές περιοχές μάλλον λίγα πράγματα. Εδώ βλέπετε την κεντρική Ευρώπη. Βλέπετε εδώ πέρα ότι κάποια πάνε καλά, αλλά ακόμα έχουμε μεγάλες διαφορές σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη. Η Πολωνία, μια χώρα η οποία μάλλον το πάει πάρα πολύ καλά με την συνοχή. Και σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2, ε, έχουμε ε, ποιοτικές ε, μετρήσεις από το 1997. Βλέπετε εδώ τη θέση μας, η οποία βελτιώθηκε και από την 44η θέση πήγε, στην, πήγε από το 44 στο 61 μάλλον. Αν όμως πάμε σε επίπεδο ΝΑΤΣ, βλέπετε ότι κάποιες περιφέρειες όπως η Μαζόβια που βελτιώσαν την ε, θέση τους, την επίδοσή τους κατά 34%. 34,4%. Και υπάρχουν κάποιες ε, άλλες που είναι κοντά σε αστικά κέντρα μεγάλα, μετροπολιτικά, ε, πάμε για 20% εκεί πέρα και στερούν κάποιες περιοχές στην Ανατολική Πολωνία κατά αυτή την περίοδο γνώσαμε μια μεταβολή 7-8-9%. Ναι. Θεωρούμε ότι το ΑΕΠ είναι ένα σωστό κριτήριο για την συνοχή και την, την πορεία του προ τη συνοχή. Τώρα, πέραν του ΑΕΠ, εδώ έχουμε διαφορετικούς δείκτες, διαφορετικά κριτήρια τα οποία προτείνονται από την πέμπτη έκθεση για την συνοχή. Δεν θα σας τα διαβάσω. Αλλά έχουμε αυτούς τους δείκτες οι οποίοι έχουν προταθεί για το ΝΑΤΣ 2. Ε, οπότε εδώ προσφέρει και ενδιαφέρον το ότι έχουμε εδώ μια καινούργια κατηγορία κριτηρίων. Τόσο μέχρι τώρα αυτά έχουν συμβαθεί για τις χώρες. Και τώρα εδώ μπορείτε να δείτε την σημασία αυτών των ε, ε, στόχων που έχουν προταθεί στα πλαίσια της πολιτικής του 2020. Έχουμε 8 κριτήρια εδώ, αντί 5. Αυτά τα προτινόμενα επίπεδα στόχους για τις χώρες αλλά και για το σύνολο της Ένωσης. Αριστερά βλέπετε τον χάρτη που λέει για την ε, ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και δεξιά το δίκτυο, το κριτήριο της παινίας που υπάρχει και εδώ βλέπετε κυρίως προς ενδιαφέρον η δεύτερη στήλη. Και λέει εδώ πέρα για την ηλικία, τα χρόνια, της ε, ικανοποίησης, της απόλαυσης της ζωής. Δανία, Φιλανδία, πάνω πάνω, 47 στη Σλοβακία. Βουλγαρία, 37. Επομένως υπάρχει εδώ μια μεγάλη διαφορά, μεγάλο χάσμα όσον αφορά την ε, ευημερία και το πόσο μακρόβι, πόσο μάλλον ζουν έχοντας την υγεία τους ο κόσμος. Βλέπετε εδώ το, αυτό το χάρτη που αφορά το ΝΑΤΣ 3 και βλέπετε ότι στα ανατολικά σύνορα έχουμε πάρα πολύ περιορισμένη προσβασιμότητα, το κάτι το οποίο επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη. Εδώ βλέπουμε την παραγωγικότητα στην τομέα τη βιομηχανία και των υπηρεσιών και εδώ υπάρχει μεγάλη διαφορά, χάσμα μεταξύ βορρά, ε, νότου, ανατολή, δύση. Εδώ ενδιαφέρον και αυτός ο χάρτη που αφορά όλες τις εκδοχές της εκδοχής α, της, ε, της έκθεσης μόνο για τη συνοχή αλλά δεν, δεν μπήκε στο τελικό κείμενο ε, μήπως σε κάποιον δεν άρεσε γιατί εδώ φαίνεται ότι έχουμε ψηλή ποιότητα διακυβέρνηση στην ε, Βόρεια Ευρώπη ε, σε σχέση με την Ανατολική Ευρώπη βλέπετε και στην Νότια Ευρώπη Νότια Ιταλία ή την Ελλάδα ή τη Βουλγαρία δεν τα πάνε καλά η Πολωνία επίσης είναι στην τέταρτη κατηγορία και πέμπτη ανάλογα με την περιφέρεια εδώ έχουμε την, την σύνδεση ή τις ευρυζωνικές συνδέσεις αναχώρα και εδώ υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Εδώ βλέπετε ε, την ανταγωνιστικότητα ως κριτήριο και εδώ μπορείτε να διαπιστώσετε ότι και εδώ έχουμε μεγάλες διαφορές ανάλογα με την περιφέρεια ε, ακόμα και μέσα στην διαχώρα Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα πόσο μεγάλη είναι η διαφορά να χάσμα χωρίζει παλιά από νέα κρατημέλη. Ποια μπορούν τα συμπεράσματα, ότι το ΑΕΠ παραμένει παρά σημαντικό κριτήριο, αλλά θα πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο υπολογισμού, τη μεθοδολογία του υπολογισμού. Πάρα πολύ σημαντικό είναι το ότι πριν από τρεις εβδομάδες πήραμε τα στοιχεία ε, για το ΝΑΤΣ 2, για το ΕΠΙΟ το 2009 και σε μερικέ χώρε ακόμα δεν έχουμε τα στοιχεία. Επομένω έχουμε μείνει πίσω πολύ. Και έχουμε κάποια ιστορικά στοιχεία με τα οποία επεξεργαζόμαστε το πρόβλημα. Δεύτερον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη διαφορετικούς συνθετικούς δείκτες, ιδίως το επίπεδο ευημερίας, και για τις περιφέρειες. Γιατί εκεί ακόμα έχουμε μείνει πίσω. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη προσοχή την κοινωνική και εδαφική διάσταση της συνοχής. Και να βελτιώσουμε την αντίληψή μας για αυτήν την διάσταση της συνοχής αυτή την πτυχή τη συνοχή, επίση θα πρέπει να δεχθούμε το ότι υπάρχει πεπρασμένο αριθμό ε, τομεακών δικτών. Σα ευχαριστώ. Thank you ε, very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στον κύριο Φρανκ Σότου, που είναι καθηγητής του Εθνικού Κέντρου ε, Τεχνών και Επαγγελμάτων και θα μας μιλήσει για τους δείκτες της πολιτικής συνοχής. Θα μας μιλήσετε για το πώς μπορεί να είμαστε ή ρεαλιστές ή συγκεκριμένοι ή και, τα δύο, ή τα δύο μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να παρουσιάσω τους ε, δείκτες του ΑΕΠ. Όλοι μισούν ε, τα οικονομικά στοιχεία, αλλά όλοι τα χρησιμοποιούν. Θα προσπαθήσω λοιπόν να επιστρέψω στα βασικά και να σας δείξω αν είναι πράγματι ρεαλιστικό να χρησιμοποιούμε ως δείκτη το ΑΕΠ. Όπως βλέπουμε σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια, ε, προσπαθούμε να πιάσουμε μια τεράστια πεταλούδα που είναι το ΑΕΠ με μικρό δίχτυ. Έχουμε πολύ μικρό προπολογισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν, ε, θέλει κανείς, αν υπόσχεται κανείς ε, ΑΕΠ πρέπει να πετύχει ΑΕΠ. Υπάρχει λοιπόν και το θέμα του ε, ότι είμαστε υπόλογοι. Μπορεί να θεωρηθούμε υπόλογοι για τα θέματα του ΑΕΠ. Η εντύπωση μου είναι ότι η ΑΕΠ, αλλά η Κομισιόν αλλάζει λίγο την άποψή τη. Μέχρι τώρα έδινε πολλά για το θέμα των δικτών επιπτώσεων. Αυτό ενδιαφέρει στο παρελθόν. Τώρα λέει η Κομισιόν, ας είμαστε πιο ρεαλιστές, ας προσπαθούμε να σκεφτούμε τα αποτελέσματα και τις, την παραγωγή και να περιορίσουμε το, τα αποτελέσματα. Και μιλάμε για περιορισμένα απο, ε, ε επιπτώσεις. Μιλάμε για καθαρά αποτελέσματα. Καθαρά αποτελέσματα, net results. Έτσι αλλάζουν τα πράγματα και κοιτάμε το θέμα των δικτών με πιο ρεαλιστικό τρόπο. Έπειτα υπάρχει το τρόπο των... Ε, κινήτρων. Υπάρχει η ανάπτυξη και η συνοχή. Μέχρι το, ε, από το 2000 ε, η έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη. Συνέχεια για ανάπτυξη μιλάμε. Ε, αλλά πρέπει να δούμε και, το, και τον τόπο των προσπαθειών. Όσο περισσότερο δίνουμε έμφαση στην ανάπτυξη, τόσο έμφαση δίνουμε στην έρευνα και ανάπτυξη. Και έκανα και τη συζήτηση με τον κύριο Μπάρκα. Δεν υπάρχουν ε, πανεπιστήμια, δεν υπάρχει τρόπος απορρόφησης της, κοινοτομίας και... και θα πάνε... πρέπει να χρησιμοποιηθεί το κοινωνικό ταμείο. Χρειάζεται απορρόφηση της έρευνας και ανάπτυξης. Οι μελέτες έχουν, έχουν δείξει αυτό. Τι κάνουμε λοιπόν. Πρέπει να φτάσουμε και στα πλουσιότερα και στα πιο αδύναμα μέρη. Δεν υπάρχουν όροι εδαφική για τους δικαιούχους. Είσαι ένα πλούσιο πανεπιστήμιο σε μια πλούσια περιοχή, μπορείς να, πά, πάρεις πολλά χρήματα χωρίς κανέναν όρο εδαφικό, χωρίς καμία ε, υποχρέωση να συνεργαστείς με τα πιο αδύναμα μέρη. Παίρνουμε λοιπόν από τους, στους, πλούσιους, και τους δίνουμε τους πόρους αυτούς και μετά ε, για τους στοχούς χρησιμοποιούμε το κοινωνικό ταμείο. My feeling is that maybe something is forgotten Και αυτό που μας αφορά είναι η εισαγωγή ορισμένων ε, τυχών. Άλλοι λένε να αφήσουμε το ΑΕΠ, ας δούμε την ποιότητα ζωής. Η ποιότητα ζωής είναι αυτή η εικόνα που βλέπετε. Βάζετε χρήματα στη στέγη, στην εκπαίδευση, στην υγεία και στο τέλος τι φτάνετε. Φτάνετε στη ποιότητα ζωής. Άρα θα πρέπει να παραμείνουμε ε, πιο απλοί. Ίσως θα πρέπει όμως να μην υπεραπλουστεύουμε, να είμαστε ρεαλιστές και όσο αφορά την λογοδοσία, ίσως το ΑΕΠ και η ποιότητα ζωής είναι δείκτες συμφραζομένων περισσότερο, δηλαδή δεν αφορούν την παρέμβαση, την πραγματική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα ας βρούμε δείκτες άμεσους που θέλουμε να δούμε σε επίπεδο κοινοβουλίου. Τι δείκτες επιθυμείτε στις εταιρικές συμβάσεις, γιατί αν δούμε το σχέδιο κανονισμού βλέπουμε ότι έχουμε έναν μακρύ κατάλογο κοινών δικτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι κοινοί δείκτες. Πώς συνδέονται με το ΑΕΠ και πώς θα χρησιμοποιηθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσαμε για τις μακροπεριφέρειες και τον τρόπο αποτίμησης. Εάν δούμε λοιπόν τα προγράμματα συνεργασίας, βλέπετε ότι υπάρχουν πολλοί δείκτες κλειδιά. Έχουμε λοιπόν μια σωρία σχεδίων και προγραμμάτων και μετά πρέπει να σκεφτείτε το ΑΕΠ. Δηλαδή, ποια είναι η συνδεσιμότητα του ΑΕΠ με αυτά τα projects, ποιοι είναι οι βασικοί δείκτες και ποιους θέλουμε να έχουμε σε επίπεδο κοινοβουλίου. Ίσως ο αριθμός προγραμμάτων δεν είναι ο καλύτερος δείκτης, όμως η κοινή δίκ αυτές ε, δεν συνδέονται άμεσα με το ΑΕΠ και δεν είναι σαφές ε, ποιοι είναι οι βασικοί δείκτες μέσα στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Ποιο είναι το πιο ε, σοβαρό, αρνητικό ή θετικό ως προς αυτές, αυτούς τους δείκτες. Ίσως, να, ίσως δεν είναι σκόπιμο να υπάρχει συνδεσιμότητα. Τι μπορούμε, πού μπορούμε να φτάσουμε τι μπορούμε να εξασφαλίσουμε, ίσως όχι το ΑΕΠ άμεσα. Υπάρχουν πολλοί δείκτες, αλλά μπορούμε να συνδεθούμε με ορισμένα ευρωπαϊκά δίκτυα, δίκτυα ε, γνώση, πλούτος, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει συνδεσιμότητα. Μία Ιταλική περίπτωση, Ιταλική περίπτωση ήταν ενδιαφέρουσα, δηλαδή ποιοι είναι οι βασικοί δείκτες, ποια είναι η προσβασιμότητα σε αυτή τη διάσταση που μπορούμε να εγγυηθούμε για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ας πούμε ότι προσπαθούμε να βρούμε έναν άλλο δίκτυ πέρα από το ΕΠ. Έναν ε, δίκτυ B για την ευρυζωνικότητα. Όλοι θέλουμε να συνδέομαστε με την ευρυζωνικότητα. Ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει κάτι το συγκεκριμένο περί αυτού. Χρειαζόμαστε την ενέργεια Ξέρουμε ότι υπάρχει χαμηλότερη παραγωγή ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι μπορούμε να κάνουμε με τα δίκτυα, τι μπορούμε να κάνουμε για τις μεταφορές. Ο κύριος Μπάρκα μας μίλησε για την καλύτερη προσβασιμότητα και στις οδικές αρτηρίες και στις σιδηροδρομικές. Αναφέρθηκε και στα αεροπλάνα, αεροπορικές μεταφορές. Ποιο είναι καλύτερος τρόπος ας πούμε για να πάμε στη Σόφια. Μπορούν όλοι οι πολίτες να έχουν προσβασιμότητα σε όλα τα δίκτυα. Ίσως η προσβασιμότητα να μην είναι το καλύτερο. Μπορούμε να σκεφτούμε και την κατάρτιση, την εκπαίδευση, ε, την διαβίου κατάρτιση, τη διαβίου εκπαίδευση, γιατί ε, τι θα κάνουμε και για αυτό το τομέα απασχόληση, απασχολησιμότητα. Υπάρχουν και άλλες διαστάσεις. Εάν θέλουμε όμως να αμφισβητήσουμε το ΕΠ θα πρέπει να βρούμε κάτι απλό. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Ε, ναι, πολύ προκλητική αυτή η παρουσίαση. Θα ανακύψουν και πολλές ερωτήσεις. Τώρα περνάμε στον κύριο Άτικάινεν. Περνάμε στη Φιλανδία. Ε, Περνάμε στον κύριο Ατικάνεν από το Ελσίν και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα υπεραπλουστεύσω τα πράγματα παρότι θεωρώ ότι δεν έχω τη δυνατότητα, είμαι δίπλα σε καθηγητές Είμαι ειδικό στη χρήση στατιστικών στοιχείων. Ασχολούμαι με εθνικές πολιτικές και σκέφτομαι, έχω μελετήσει το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Με τα μεγάλη μου χαρά θα σας παρουσιάσω κάποιες ιδέες για τον οποίο μπορούμε να μετρήσουμε την συνοχή και θα πω και λίγα πράγματα για την ανταγωνιστικότητα. Θα θυμόσαστε τη δεύτερη διαφάνεια του καθηγητή Σωτός, όπου υπάρχει ανάπτυξη και συνοχή. Εγώ τα πράγματα τα βλέπω αντίστροφα. Εγώ θεωρώ ότι οι δρόμοι αυτοί οδηγούν στον ίδιο στόχο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι η ισχυρή αναπτυξιακή πολιτική είναι καλύτερη πολιτική συνοχής αν μετράμε την ε, συνοχή πρέπει να μετράμε και την ανταγωνιστικότητα των περιοχών και η δομή του περιφερειακού συστήματος είναι βασικό στοιχείο. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να υπογραμμιστούν τα δημογραφικά στοιχεία και επίσης ότι όλα τα μέτρα θα πρέπει να έχουν σχέση με την πολιτική και να ε, λαμβάνουν υπόψη τους την κλίμακα. Τώρα θα υπεραπλουστεύσω. Αν σκεφτούμε την περιφερειακή, τους δείκτες περιφερειακής ανάπτυξης, έχουμε το ΑΕΠ με τους περιορισμούς που ήδη ακούσατε, κάτι άλλο που προσπαθούμε να μετρήσουμε και να παρακολουθήσουμε είναι η θέση εργασίας, ε, απασχόληση, ανεργία. Και τρίτον, τα δημογραφικά στοιχεία οι μορφές μετανάστευσης είναι αυτές που παρακολουθούμε γιατί είναι ο ταχύτερος δείκτης για τις περιφερειακές επιδόσεις. Όλα αυτά είναι τα παραδοσιακά που γνωρίζουμε από τις δεκαετίες του 50 και του 70. Αυτό το τρίγωνο. Το βασικό κρίσιμο ζήτημα εδώ που ε, συχνά αναφέρεται είναι να βρεθεί η γωνία της αρμοδιότητας, της δεξι... Ε, ικανότητας πώς θα πρέπει να, μετρεύε, να μετρείται αυτή. Πρέπει να, δώσουμε περισσότερο ενδιαφέρον, να δείξουμε περισσότερο ενδιαφέρον γι' αυτό. Και βεβαίως το θέμα της πολιτικής είναι ζωτικής σημασίας. Προσπαθούμε να πετύχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη, ολοκληρωμένη ανάπτυξη που θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της όλη την ε, κατάσταση των πολιτών ολοκληρωμένα και πολύ χάρηκα που το είδα αυτό σε πολλές διαφάνειες, να και άλλη μία η σχέση ανάμεσα στο ΑΕΠ και την ποιότητα ζωής. Εδώ βλέπετε το ΑΕΠ και την γενική ικανοποίηση από τη ζωή. Βλέπετε ότι το ΑΕΠ ανεβαίνει αλλά δεν αφορά καθόλου ε, την γενική ικανοποίηση με τη ζωή. Προφανώς λοιπόν έχουμε κάποια κενά πληροφόρησης ε, για την μέτρηση των περιφερειακών επιδόσεων. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια ολιστική αντίληψη, κάτι που το δουλεύει η Eurostat και είναι πολύ σημαντικό ζήτημα. Μετράτε το περιβάλλον κλπ. Και επίσης το πόσο ευάλωτο είναι το σύστημα στις εξωτερικές, στα εξωτερικά χτυπήματα. Και τέλος θα μιλήσω για, την, για τις πολλαπλές κλίμακες και τα θέματα ηλικίας και πληθυσμού. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα ε, ενός σύνθετου δίκτυ που περιλαμβάνει και το ΑΕΠ και την απασχόληση και την έρευνα και ανάπτυξη. Το δημιούργησε ο Τόμας Χανέλ από τη Φιλανδία, το Eurofutures. Futures είναι αρκετά γνωστή η εικόνα των πιο ανταγωνιστικών περιοφεριών της Ευρώπης. Όμως υπάρχει και το θέμα της κλίμακας και πρέπει να το μάθουμε. Ξέρω ένα μέρος από την Ανατολική Φιλανδία. Αν δείτε πάνω δεξιά στη Φιλανδία, βλέπετε ότι εκεί δεν πάει πολύ καλά η κατάσταση. Είναι στο χαμηλό τεταρτημόριο. Και αν δείτε από το επίπεδο ΝΑΤΣ 2 στο ΝΑΤΣ 3, θα δείτε ότι δεν υπάρχει ε, κάποιος κινητήρας που να βλέπουμε στο επίπεδο νατς 3. Στο νατς 4 όμως βλέπουμε την πατρίδα ενός μέλους εδώ της αίθουσας, του, το Βάρτακας, που είναι μια ισχυρή βιομηχανική περιοχή και λίγο παραπάνω από εκεί υπάρχει το Κουόπιο που είναι κέντρο ε, ικανότητας ε, της Ανατολικής Φιλανδίας. Και εκεί που ε, αν πέσει το Κουόπιο είναι πολύ θα πέσει και όλη η Ανατολική Φιλανδία και άρα πρέπει να ξέρουμε πόσο καλά ε, λειτουργεί αυτός ο κινητήρας. Η δυσκολία εδώ είναι να τα συνδέσουμε όλα αυτά. Είναι το θέμα της προσβασιμότητας. Ε, η απόσταση είναι περίπου 70 χιλιόμετρα ανάμεσα στα δύο αυτά μέρη. Αλλά υπάρχουν ε, κάποιοι κόμβοι μικροί και μεγάλοι που πρέπει να συνδυάζονται εντός των περιφερειών και ε, στο κράτος και στην Ευρώπη και παγκόσμια. Υπάρχει και το δημογραφικό ζήτημα. Εδώ βλέπετε τον πληθυσμό ηλικίας άνω των 65. Εδώ βλέπετε μια παρόμοια εικόνα σε επίπεδο ΝΑΤΣ 3. Θα σας δείξω όμως γιατί ενδιαφέρεται για το θέμα η Φιλανδία. Εδώ βλέπετε ότι οι μπλε γραμμές είναι περιοχές ΝΑΤΣ 2 και δείχνει το 2020. Η κόκκινη γραμμή είναι ο εθνικός μέσος όρος. Η Φιλανδία τώρα αντιμετωπίζει το πρόβλημα της δημογραφία, αλλά υπάρχει και η Ιταλία, η Γερμανία και η Γαλλία που και εκεί ε, αυξάνει ο μέσος όρος ηλικίας και ε, το θέμα αυτό θα μας αφορά σε ερχόμενες ε, δεκαετίες. Τέλος. Αυτό που μετράμε επηρεάζει αυτό που κάνουμε και αν οι μετρήσεις μας είναι σφαλμένες, ίσως υπάρχει στρέβλωση και στις αποφάσεις και θα είναι αποφα... παίρνουμε αποφάσεις που δεν θέλαμε να πάρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε τώρα θα αρχίσει η συζήτηση. Α, έχουμε άλλον έναν ομιλητή. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη. Ναι, από το ε, Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βελγίου, ε, το ULB. Βεβαίως. Ε, Θα ήθελα συνοπτικά να σας μιλήσω για τα αποτελέσματα μιας μελέτης που μας ζητήθηκε και αυτό που μας απασχολεί είναι κατά πόσο μπορούμε να βρούμε έναν καλότερο δείκτη από το ΑΕΠ και από τον ε, περιφερειακό εθνικό δείκτη για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε έναν απλό δείκτη και από την άλλη πλευρά να χρησιμοποιήσουμε αξιόπιστα δεδομένα από πλευράς Eurostat. Για να επανέλθω στο θέμα που ήδη εφήγει από τους προλαλήσαντες, θα ήθελα να πω ότι το ΑΕΠ θέτει ε, γνωστικά προβλήματα, ε, θέματα συλλογιστικής και τρόπου σκέψης. Όταν το χρησιμοποιούμε για την οικονομική συγκυρία δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως όταν χρησιμοποιείται ως διαρθρωτικός δείκτης υφίστανται προβλήματα διότι η αύξηση του ΑΕΠ μπορεί να προέρχεται ε, από την αύξηση της παραγωγής η οποία κοινωνικά είναι άχρηστη. Το ζήτημα όμως που τίθεται είναι κατά πόσο μπορούμε να ε, προσαρμόσουμε το ΑΕΠ σε έναν περιφερειακό ακαθάριστο δίκτυ για να μετράμε τα περιφερειακά αποτελέσματα. Από θεωρητικής πλευράς, μία από τις μεγάλες δυσκολίες είναι η εξής. Θα θέλαμε η οικονομική ανάπτυξη να αφορά την εθνική επικράτεια ή θέλουμε να βελτιστοποιήσουμε παντού το επίπεδο ζωής του πληθυσμού. Αυτό είναι κάτι το εντελώς διαφορετικά. Δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι σε ορισμένες περιφέρειες θα μπορούσαμε να έχουμε μία ευημερία η οποία να συνδέεται με κάτι άλλο από την περιφερειακή παραγωγή. Εάν λοιπόν φτάσουμε στο θέμα των ε, τεχνικών δυσχεριών για το περιφερειακό ΑΕΠ, υπάρχει το θέμα των συνόλων των εθνικών ΑΕΠ, των ΑΕΠ της επικράτειας σε περιφερειακό επίπεδο. Εάν λάβουμε υπόψη την προστιθέμενη αξία που συνδέεται με τους ε, μισθούς, θα μπορούσαμε να αποδώσουμε υψηλό ΑΕΠ για μία, στα πλαίσια μιας εταιρεία ή επιχείρησης στην έδρα της και όχι στον τόπο παραγωγής. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μία συνοχή που να έχει αντίκτυπο σε όλες τις περιφέρειες. Το άλλο θέμα είναι ότι δεν έχουμε ε, δείκτες για την ε, αγοραστική δύναμη γιατί οι τιμές στο Παρίσι και στην περιοχή Λιμουζά δεν είναι οι ίδιοι. Δεν μπορούμε να μιλάμε λοιπόν για παρόμοιες τιμές. Ως προς τον κατακαιρματισμό, τον διαχωρισμό, ισχύει σε επίπεδο ΝΑΤΣ 3 αλλά και ΝΑΤΣ 2 και 1. Όλοι ξέρετε ότι οι Βρυξέλλες βρίσκονται στο ΝΑΤΣ 1 που υπάρχει υψηλό ΑΕΠ ανα, και, κατά αλλά αυτό δεν ισχύει σε άλλες περιφέρειες. Ακόμα και στην ευρύτερη περιφέρεια των Βρυξελών. Αυτές είναι σκέψεις τεχνικών δυσχεριών. Τι μπορούμε να βρούμε ως εναλλακτική λύση. Είδαμε αρκετούς ε, διαθέσιμους δείκτες και βλέπουμε ότι ε, αν ταξινομήσουμε τους δείκτες αυτούς, Υπάρχει ένας καλός συσχετισμός μεταξύ ΑΕΠ ως οικονομικού δείκτη, τους δείκτες ηλικής ευημερίας που μπορούμε να μετρήσουμε με το εισόδημα μετά από τις, ε, από τις, ε, από τις αφαιρέσεις που γίνονται για, τους, ε, για τα διάφορα ταμεία Επίσης το προσδόκιμο ζωής, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές, αναπεριφέρεια ιδιαίτερα για τους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες και επίσης το ανθρώπινο κεφάλαιο, το ποιοτικά ανθρώπινο κεφάλαιο, το οποίο ε, είναι διαφορετικό, ανάλογα και με τη χρήση των ε, τεχνολογιών επικοινωνίας. Όμως οι δείκτες είναι ευάλωτοι όταν μιλάμε για τη μακροχρόνια ανεργία, για την κατάσταση ένδυας των πολιτών και θα πρέπει να δούμε κατά πώς υπάρχει σύγχυση με τους οικονομικούς δείκτες, διότι σήμερα υπάρχουν φύλακες φτώχειας σε πολύ μεγάλες, σε μεγάλες πόλεις οι οποίες ευημερούν. Άρα εδώ οι συσχετισμοί είναι αρνητικοί. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη αυτές τις κοινωνικές αποκλίσεις, αλλά δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με τους οικονομικούς δείκτες. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, το οποίο χρήζει άλλων κριτηρίων. Ως προς τους περιβαλλοντικούς δείκτες, δεν τους βλέπετε στον πίνακα αυτό, στους πίνακες αυτούς, γιατί είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν σε περιφερειακό επίπεδο. Άρα είναι καλύτερα να επικεντρωθούμε, να επικεντρώσουμε όλους τους δείκτες μόλυνσης σε περιφέρειες ή πρέπει να γίνει ε, ομοιογενής κατανομή στην επικράτεια. Αυτό το θέμα δεν έχει επιληθεί και άρα το περιβαλλοντικό ζήτημα θα πρέπει να μας απασχολήσει κάπως διαφορετικά με διαφορετικούς δείκτες και διαφορετικό τρόπο σκέψης από τους, ε, σε σχέση με τους οικονομικούς δείκτες. Επειδή έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, ε, θα ήθελα να πω ότι έχουμε μία θεωρητική επιλεξιμότητα των περιφερειών με βάση το κατόφλι του 75% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και όχι 90% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ε, έχετε το ΑΕΠ αριστερά και ένα ΑΕΠ συν δεξιά λαμβάνοντας υπόψη τα, ε, τα καθαρά εισοδήματα, το καθαρό εισόδημα. Το ίδιο έγινε με ένα ΑΕΠ συν 3 λαμβάνοντας υπόψη δηλαδή την υγεία και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε ποια είναι τα τελικά αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μερικές περιφέρειες της Δυτικής Ευρώπης χάνουν την επιλεξιμότητά τους γιατί έχουν πολύ υψηλές κρατήσεις, κοινωνικές κρατήσεις και για τον τομέα της πρόνοιας. Υπάρχει γύρανση του ε, πληθυσμού που επιστρέφει στον ε, τόπο προέλευσης μετά τη σταδιοδρομία. Εδώ λαμβάνω υπόψη το, την περιοχή του Λιμουζά. όπου με βάση αυτές τις ε, κοινωνικές μεταφορές υπάρχει εξισορρόπηση, ενώ στις ανατολικές περιφέρειες η πρωτεύουσα είναι επιλέξιμη όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν μεταφορές κοινωνικών δικτών σε, στο υπόλοιπο της χώρας, αλλά παρόλα αυτά αυξάνεται η επιλεξιμότητα της πρωτεύουσα. Αυτός είναι ο τελικός χάρτης όταν βλέπουμε το ΑΕΠ και την υγεία και το ανθρώπινο δυναμικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο Βλέπετε όμως ότι υπάρχει μία επιβάρυνση, γιατί βλέπουμε όποιο και να είναι το επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών, θα πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής ευαλωτότητας. Και αυτό αφορά περιφέρειες οι οποίες ευημερούν σε οικονομικό επίπεδο. Ευχαριστούμε τον καθηγητή Βάντερ Μάτεν. Θα ήθελα και η Κομισιόν να λάβει το λόγο. Ίσως, Ίσως ε, προς το τέλος της ζήτησε να λάβετε το λόγο. Εδώ τώρα ποιοι να το λόγο. Πρώτος ο Γιάννη Άλμπρεχτ. Ναι, σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον εμείς ε, ως ε, πολιτικοί να ακούμε τους αναλυτές αυτών των στατιστικών κλπ. Θυμάμαι κάπου, κάποτε με ρώτησαμε ποιο είναι το ΑΕΠ και είπε 74. Τέλος πάντων θα μπορούσαμε να πάμε για καλύτερα και, άλλα, και άρα οι στατιστικές είναι μεταβλητές. Για την ανάπτυξη τώρα. Ναι. Πιο πλούσιοι επενδύον Το 7ο, το 6ο και το 5ο πρόγραμμα. Τα προγράμματα τα ίδια λένε. Τώρα είναι το θέμα της αριστείας, να αποφύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Εάν θέλουμε να βοηθήσουμε την Ευρώπη να αναπτυχθεί, θα πρέπει να επενδύσουμε στις περιφέρειες. Έχουμε δύο πραγματικότητες όμως να αντιμετωπίσουμε. Η πρώτη είναι πώς ορίζεται, πώς περιγράφεται ο ρυθμός της ανάπτυξης, το ειδικό επίπεδο κλπ. κλπ. Και έχουμε μια ποικιλία κριτηρίων. Και αυτό είναι και το ενδιαφέρον. Και κατόπιν έρχεται η ώρα των πολιτικών αποφάσεων, που πάντοτε είναι το κατακεφαλήν εισόδημα. Το επ κατακεφαλήν. Άρα το που πάνε οι πόροι είναι θέμα ΕΠ. Κατόπιν έχουμε την αξιολόγηση των πολιτικών. Αποτελεσματικότητα κλπ. Το πώς θα μετρήσουμε, το πόσο αποτελεσματική είναι μια πολιτική. Έχουμε διαφορετικά κριτήρια, δείκτες για την αποτελεσματικότητα και κατόπιν έχουμε τα κριτήρια του πού θα πάνε τα τι είναι επιλέξιμη και κατόπιν έχουμε το Το Άρα θα πρέπει να ρίξουμε ματιά σε όλους τους χάρτες και βλέπουμε ότι οι διαφορές παραμένουν. Ίδια κατάσταση. Και ίσως δεν θέλουν κάποιοι να δείξουν την πραγματικότητα γιατί θα πάψουν να επιλέξουν και να τους κυνηγήσουν οι ψηφοφόροι. Άρα, θα πρέπει να αποτυπώνεται κάπως έτσι η κατάσταση για να, για να προβληματίζονται οι πολιτικοί εμείς ή θα πρέπει ή να, να θεωρήσουμε ότι δεν, αντιμετωπίζει, δεν, δεν αποτυπώνεται έτσι η πραγματικότητα. Είναι περίπλοκη κατάσταση, αλλά αυτό αφορά και την αξιολόγηση αποτελεσματικότητα, αλλά αφορά και την απόφαση του ποιο είναι επιλέξιμος. Ιδάλλως, θα είμαστε σε μια σχιζοφρενική κατάσταση. Άλλα θα μετράμε και άλλα μέτρα θα λαμβάνουμε. Ίσως κάποια στιγμή ο χάρτης θα δείξει ότι οι πιο ευτυχισμένοι αυτοί που έχουν το χαμηλότερο ΑΕΠ. Άρα, πού θα πάνε τα χρήματα, στους πιο πλούσιους στους πιο ευτυχισμένους ή στους λιγότερο ευτυχισμένους. Φανίστερο. Και κατόπιν θα απαντήσουν ε, οι προσκεκλημένοι μας. Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτά στη διάθεσή μας και μπορούμε να τα συνδυάσουμε, να τα συνθέσουμε αλλά λάβουμε όλα αυτά που ακούσαμε υπόψη και επομένω αξιόλογα αυτά τα οποία ακούσαμε ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη, αλλά το ΑΕΠ καθε αυτό παραμένει πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο για την ανάπτυξη. Όταν κατανέμονται κάποιοι πόροι, είναι δυνατόν να ληφθούν υπόψη και άλλα κριτήρια, αλλά δεν μπορεί κανείς να αφήσει στην άκρη το ΑΕΠ που είναι τόσο σημαντικό, σημαντική υπόθεση. Και το πόσο θα πετύχει μια πολιτική, ας πούμε, στρατηγική του 2020, ε, μας, μας έδωσε κάποια στοιχεία. Επομένως, κατόπιν το όσων ακούσαμε, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι με το ΑΕΠ συν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια κριτήρια που έχουμε σήμερα. Έχουμε δεδομένα τόσο ποιοτικά που να μας επιτρέπουν να ενεργήσουμε έτσι. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Γιατί όταν έρχεται η ώρα να αξιολογήσουμε κάποια προγράμματα το οποίο θα γίνει στο άμεσο μέλλον, τι θα κάνετε σε σχέση με αυτό που είπα. Τώρα για την εδαφικότητα. Υπάρχει η αρχή της υποκριτικότητας. Και έτσι λαμβάνονται οι αποφάσεις για τις Βρυξέλλες και τις άλλες περιφέρειες και ασκείται η περιφερειακή πολιτική. Προσθέσαμε τώρα επομένως την εδαφικότητα. Και είναι σημαντικό αυτό. Θα πρέπει αυτό, δηλαδή η δαφικότητα, να συντεριάξει με τα υπόλοιπα στοιχεία, τα υπόλοιπα κριτήρια. Τέλος, αυτό το οποίο δεν περιέλαβε προτάσεις η Επιτροπή είναι η αριστεία για έρευνα και ανάπτυξη. Οι περιφέρειες που έχουν το στοιχείο της αριστείας. Αυτό δεν περιελήφθη στις προτάσεις. Εξήταζα, μελετούσα ότι υπάρχει σε σχέση με τη συνοχή για τα νέα κρατημέλη. Εκεί προσπαθούν να δημιουργούν κέντρα αριστείας. Αυτό παρελήφθη. Θα πρέπει να το προσέξω. Και ίσως θα πρέπει να τεθούν οι σχετικοί κανόνες για το... Σέτερ. Κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, Ελίζαβετ. Äh Καταρχήν θέλω να πω ότι χαίρομαι που οργανώσαμε αυτή τη ε, μικρή ακρόαση, παρόλο που τα περισσότερα μέλη απουσιάζουν. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να μεταβιβάσουμε τις πληροφορίες. Είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα. Μας απασχολεί από καιρό και μάθαμε πολλά. Με το ΑΕΠ διαπιστώσαμε ότι δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εδαφική και κοινωνική συνοχή. Και το ΑΕΠ είναι απλά πολύ περιορισμένο για να μας δώσει αυτές τις πληροφορίες και τα δεδομένα είναι στρεβλά και με βάση αυτά φτιάχνουμε τα καθίσματα, τους πάγκους πάνω στους οποίους καθόμαστε. Θεωρούμε ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν κάποια να, φτάσουν, να φτιάξουν, αλλά τα αποτελέσματα της Κομισιόν δεν δείχνουν κάτι τέτοιο. Διαπιστώνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι πάντα περιορισμένα. Μα γιατί, για, επειδή οι δείκτες που έχουμε στη διάθεσή μας δεν μπορούν να δώσουν την πραγματική εικόνα και τα δεδομένα είναι στρεβλά. Αυτό που ακούσαμε από την τελευταία ομιλία του κυρίου Βάντερ Μότεν το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Τη στιγμή κατά την οποία το ΑΕΠ που είναι βασικό ή εν πάση σημαντικό κριτήριο δεν λέω ότι μπορούμε να αποφασίσουμε χωρίς να στηριχθούμε στο ΑΕΠ, γιατί τα οικονομικά στοιχεία είναι σημαντικά. Αλλά αν μείνουμε μόνο σε αυτά, η κατάσταση. Κάποιες περιφέρειες εμφανίζονται πολύ καλύτερες από ό,τι είναι στην πραγματικότητα, αν τα ε, παρακολουθήσουμε λίγο πιο, από πιο κοντά, αν λάβουμε υπόψη μα και κοινωνικά κριτήρια. Γι' αυτό η, τα θέματα δεν είναι μόνο οικονομικά, είναι και κοινωνικά και εδαφικά. Κάποιες ε, αστικές αναπτύξεις ας πούμε που θε, επισήμως είναι θετικές αλλά αν τις κοιτάξουμε κοινωνικά κριτήρια διαπιστώνουμε κάτι άλλο γιατί η αύξηση του εισοδήματος αφορά λίγους μόνον και όχι την μεγάλη πλειονότητα. Πρέπει λοιπόν να έρθει, λέμε, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να τη σταθμίσει. Αν δεν στηριχτούμε μόνο στο ΑΕΠ, ε, θα καταλάβουμε γιατί υπάρχει η στασιμότητα στην ανάπτυξη, ας πούμε. Επειδή η ε, ανάπτυξη μετρήθηκε μόνο με βάση το ΑΕΠ. Αν είχε προσθεθεί και ένα άλλο κριτήριο αξιολόγησης, η εικόνα θα ήταν πολύ πιο ακριβής και θα είχαμε συνειδητοποιήσει ότι η παρέμβαση θα έπρεπε να είχε ε, γίνει και σε άλλα επίπεδα. Επίσης ε, εκτιμώ ιδιαίτερα την, αυτά που ακούσαμε για τις ε, αγροτικές περιοχές, για το εδαφικό σκέλος δηλαδή, όπου είναι απολύτως σαφές ότι το ΑΕΠ δεν εξαρτάται απευθείας ή άμεσα από την κατάσταση των περιοχών αυτών όσον αφορά την προσβασιμότητα, την, πρέπει να δούμε πώς θα ε, διαφοροποιήσουμε τα πράγματα. Επίσης έχουμε λιγότερους πόρους και στην Ανατολική και στην Κεντρική Ευρώπη. Έχουμε λιγότερους πόρους από ότι και για την Ρουμανία και Βουλγαρία. Επειδή υπάρχουν λιγότεροι πόροι, αν πρέπει να παρέμβουμε πραγματικά στοχευμένα πρέπει δίπλα στο ΑΕΠ να προσθέσουμε και άλλα κριτήρια. Προσθήκη κριτηρίων είναι το σημαντικό. Και νομίζω ότι η πρόταση του κυρίου Βαντεμόταν επ' αυτού ήταν ξεκάθαρη. Υπάρχει σοβαρή αντίφαση ανάμεσα σε αυτά που ακούσαμε από τους διάφορους ομιλητές. Ο κύριος Σράτα είπε ότι έχουμε μόνο το ΑΕΠ και τίποτα άλλο, ενώ οι άλλοι ήταν πιο σαφείς. Είπαν ότι υπάρχουν όρια ε, του ΑΕΠ, στο ΑΕΠ ως δίκτυ για να απεικονιστεί η πραγματικότητα. Στο Σλάτα, στον κύριο Σλάτα λοιπόν, πώς κρίνετε εσείς αυτά που είπαν οι συναδελφοί σας, οι οποίοι μοιάζει ότι έχουν διαφορετικές απόψεις από εσά. Αυτή είναι η βασική μου ερώτηση, όπως έχετε αντιληφθεί. Έχω όμως και άλλη μία που ε, απευθύνεται στον κύριο Βάντε και στον κύριο Σοτού. Εάν πράγματι ισχύει ότι μπορεί το ΑΕΠ να διορθωθεί με την προστίχη άλλων κριτηρίων. Υπάρχει η οικονομική ανάπτυξη βεβαίως, αλλά διαπιστώνουμε ότι αυτή αφορά μόνο κάποιο μέρος και αν το μελετήσουμε ακόμη πιο προσεκτικά θα διαπιστώσουμε ότι αφορά κάποιους λίγους ανθρώπους. Αν όλα αυτά ισχύουν, τι προτείνεται στην πράξη την οποία έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε. Το, οι περιφέρειες έχουν καταταχεί με βάση το ΑΕΠ τους, όπως προτείνει ο κανονισμός, πράγμα που σημαίνει ότι ήδη κάνουμε βασικά λάθη. Μήπως θα έπρεπε να προσθεθούν συμπληρωματικά κριτήρια στον κανονισμό για να διορθώσουμε την κατάσταση. Υπάρχουν τα ποσοστά, οι συμπληρωματικοί δείκτες, Όλα αυτά θα μας επιτρέψουν ε, να επενδύσουμε τους πόρους μας με πιο διαφορετικό τρόπο. Ποιος είναι ο συγκεκριμένους τρόπους που προτείνετε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Λέει η κυρία Ντέλη. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Νομίζω ότι δεν απαντάτε σε όλα τα ερωτήματα, διότι εδώ πολύ καιρό, πολλοί οικονομολόγοι λένε ότι το ΑΕΠ δεν θα επιλύσει το θέμα μας και δεν θα ε, ανταποκριθεί στις διεθνείς ε, και περιφερειακές ε, προκλήσεις, γιατί ζούμε σε ένα κόσμο που συνεχώς μεταλλάσσεται. Και με βάση αυτή τη διαπίστωση Νομίζω ότι εξ αρχής έχουν επινοηθεί λάθος οι δείκτες. Είναι λάθος η μεθοδολογία, αυτή η μεθοδολογία. Και ένα από τα πράγματα που υπενθυμίσαμε είναι η ανάπτυξη, ο δείκτης ανάπτυξης που μας επιτρέπει το ΑΕΠ. Όμως ο τρόπος παραγωγής και κατανάλωσης μας δείχνει ότι αν έχουμε μόνο αυτό το δείκτη δεν θα ε, προωθηθεί στο δίνεκες, όπως ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε και σε έναν και μοναδικό πλανήτη. Ξού και θα πρέπει να δούμε τις πολιτικές συνοχής. Θα πρέπει να συνδέσουμε τον τρόπο κατανάλωσης και καθώς και τα οικολογικά δεδομένα. Νομίζω ότι θέσαμε δείκτες που ε, είχαν μία αποσύνδεση μεταξύ πραγματικής οικονομίας και σκιώδους οικονομίας ή εικονικής οικονομίας με βάση τον πλούτο. Άρα, πώς ορίζουμε ως πλούτο για τις περιφέρειες, πού έγκυται ο πλούτος σε σχέση με την, το σύστημα υγείας ως προς την απασχόληση, την ανεργία και ούτω καθεξής. Αυτό το θέμα είναι ύψης της σημασίας. Δεύτερον, μας ε, λέτε ότι επί του παρόντος ε, ε, δεν έχουμε άλλες επιλογές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη διάσκεψη του Johannesburg είχε γίνει λόγος για ευημερία και μιλήσαμε και για το οικολογικό αποτύπωμα αποτύπωμα το περίφημο. Μιλήσαμε λοιπόν για παραγωγή, για κατανάλωση, για κινητικότητα, πώς ορίζεται η κινητικότητα στην υφήλιο στην επικράτεια, πώς έχει αστεί φιλία και ούτω καθεξής. Το θέμα των δικτών είναι και θέμα δημοκρατίας. Κανένας δεν ρώτησε τους Ευρωπαίους πολίτες τι μετράει στη ζωή τους για να είναι πιο ευτυχείς. Έχουμε και το ε, εγχείρημα της συμμετοχής, δηλαδή στην περιοχή Παντεκαλέ, όπου, υπήρξε μεγάλ, όπου υπήρξαν μεγάλες κινητοποιήσεις, ε, ρωτήσαμε τι σας κάνει ευτυχής η φτώχεια είναι ο πρώτος παράγοντας μη ευτυχίας, επίσης το θέμα της υγείας και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν έχει το θέμα της συμμετοχής. Θα ήθελα τώρα οι εμπειρογνώμονες να απαντήσουν, να αποφασίσουν μεταξύ τους ποιος θα λάβει το λόγο πρώτα, με την ίδια σειρά ή όχι και ούτω καθεξής. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις σας. Πρώτα-πρώτα σας παραπέμπω στα συμπεράσματά μου. Γιατί ίσως κάποιοι βουλευτές δεν καταλαβαίνουν καλά, ίσως γιατί δεν τα είπα με αρκετή σαφήνεια. Είπαν ότι το ΕΠ είναι σημαντικό κριτήριο, θα πρέπει να βελτιώσουμε την αθολογία των υπολογισμών. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το ΑΕΠ καθε αυτό. Ακούσαμε πολλά όσον αφορά την σύγκριση σε περιφερειακό επίπεδο και είπαμε ότι κάποιες μητροπολιτικές περιοχές έχουν πάρα πολύ ψηλό ΑΕΠ και κυρίως οι πρωτεύουσες. Δεν υπολογίζουμε σωστά την παραγωγή εκτός αυτών των περιφερειών. Φασοβία, Πράγα εννοώ, Βουδαπέστη. Ούτε τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τις περιλαμβάνουμε. Να, ένα άλλο παράδειγμα. Βλέπετε πόσο επιδέχεται βελτίωση το τι κάνουμε. Ήδη είπαμε ότι υπολογίζουμε την παραγωγή που βλάπτει το περιβάλλον. Και υπάρχουν πολλοί λόγοι που μας οδηγούν στην βελτίωση της μεθοδολογίας μας και στο μισό της εγγύσης μας σας είπα ότι θα πρέπει να δούμε τους συνθετικούς δείκτες. Δηλαδή το επίπεδο ευημερίας σε σχέση με τον πλούτο των εθνών η Eurostat και οι εθνικές αστικές υπηρεσίες. Αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Με κάποια έθνη, κράτη ή τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. θα πρέπει εδώ να λάβουμε υπόψη και την ταφική ε, και κοινωνική πτυχή και δεν όπως τον Γιάνν Άλμπριχτ ότι είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπε Ναι, χρησιμοποιούμε αυτά που λέει η συνθήκη. Κοινωνική, οικονομική, εδαφική πτυχή και από αυτού προσπαθούμε να δαπανίσουμε ορθολογικά τους οικονομικούς πόρους. Έχουμε όμως και την πολιτιστική συνοχή και την πολιτική συνοχή της Ευρώπης. Και αν αυτές τις ε, πτυχές τις ε, λάβουμε υπόψη, τότε το πού θα πάνε οι οικονομικοί πόροι είναι επίσης σημαντικό και έτσι θα διακυβευτεί το αν θα βοηθήσουμε την ανάπτυξη. Τι λείπει από το σχέδιο ή τα σχέδια κανονισμών. Έχουμε κάποιους πάρα πολύ γενικούς δείκτες και κριτήρια για κάποια προγράμματα και κατόπιν κάποιους λειτουργικούς επιχειρησιακούς πόσοι συμμετέχουν, πόσε επιχειρήσει και επίσης και το ΑΕΠ. Και λέτε, εσείς που είστε δική να σας τα εξηγήσουμε, λέτε. Μα θα πρέπει να δούμε τους συγκεκριμένου στόχου σε ενωσιακό επίπεδο. Συγκεκριμένοι δείχτες. Και θα πρέπει κανείς να δει σαν δεδομένα τις κινήσεις που γίνονται, τις δράσεις, είναι πάρα πολλές. Προσβασιμότητα είναι και αυτό ένας δείκτης. Τα έχουμε συζητήσει, αλλά δεν έχουμε δει τι γίνεται σε ενωσιακό επίπεδο. Έναν δείκτη προσβασιμότητος που να μην το συνδέσουμε με την ανάπτυξη. Για να υπάρχει ανάπτυξη θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα στην ανάπτυξη. Μια δίκαιη δίκαιος βαθμός προσβασιμότητας. Η προσβασιμότητα επομένω είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ um, Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Αυτό κάνουν όλες οι χώρες, παίζουν με τα όρια και τους κανόνες και μας εκπλήσει πάντα το ότι δεν έχουμε κανόνες που να είναι σαφές ότι θέλει κανείς να ξεπεράσει τα όρια, να έχει κάποια ανταμοιβή για την προσέγγιση ότι εγώ θα είμαι καλός. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες πρέπει κανείς να ξεπεράσει κάποια όρια. Υπάρχουν απ' την άλλη άλλα προγράμματα όπου οι περιφέρειες δεν έχουν ενδιαφέρον να, ή συμφέρον να ξεπεράσουν τα όρια. Το ξεπέρασμα των ορίων ε, πρέπει να προσφέρει ανταμοιβή. Θέλω να απαντήσω σε αυτό το θέμα για το εδαφικό επίπεδο. Το αστικό σύστημα διαφέρει από χώρα σε χώρα. Όπως έδειξα στην ε, Φιλανδία έχουμε τέσσερα τέτοια επίπεδα. Ε, χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση ε, των βασικών μονάδων της καθημερινής ζωής στην Ευρώπη. Τέλος, θέλω να πω ότι ε, συμφωνώ ότι πρέπει να συμπεριληφθούν και να προχθούν οι περιφέρειες ε, υπεροχής είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε και να μετρήσουμε το επίπεδο ικανότητας και τις ροές και, των σχέσ, και τις σχέσεις ανάμεσα σε αυτούς τους κόμβους ε, απόδοσης. Για να απαντήσω στην τελευταία παρέμβαση, Γνωρίζω ότι το, πολύ καλά ότι το ΑΕΠ δεν είναι ο καλύτερος δείκτης για να ανταποκριθούμε στις διεθνείς προκλήσεις και για την αηφόρο ανάπτυξη. Όμως το εγχείρημα αυτό αφορά μία απλούστευση του εγχειρήματος και του ότι τοποθετούμε σε μια προοπτική κατανομής και προσαρμογής των κριτηρίων συνοχής. Άρα παραμείναμε σε αυτό το πλαίσιο. Βεβαίως, ε, τι θα πρότεινα, ως προς το τι θα πρότεινα να προσθεθεί στο ΑΕΠ, μα το προείπα. Έναν δίκτυ ευημερίας και Ίσως θα πρέπει να λάβουμε τα, τα καθαρά έσοδα και όχι τα καθάριστα. Ίσως είναι η καλύτερη λύση. Ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, μάλλον αυτό, ένας δείκτης που οδηγεί σε διακρίσεις είναι το προσδόκιμο ζωής των ανδρών, που διαφέρει από των γυναικών, καθώς και τα κριτήρια κατάρτισης και εκπαίδευσης. Θα πρέπει λοιπόν η Eurostat να μας δώσει αριθμητικά στοιχεία έρευνας και ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο που να είναι καλύτερα από αυτά που διαθέτουμε έτσι ώστε να έχουμε όχι μόνο εθνικές ποσοστιαίες αναλογίες αλλά στοιχεία σε επίπεδο NATS 2 για να μπορέσουμε να προβούμε στη βελτίωση των δικτών. Επίσης θα ήθελα να εξετάσουμε την κατανομή που ισχύει σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2 και 3 και να το προσαρμόσουμε σε επίπεδο απασχολησιμότητας, δηλαδή τόπου εργασίας. Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχουν κατανομές σε επίπεδο ΝΑΤΣ 2 και ΝΑΤΣ 3, ενώ στο Βέλγιο που έχει ομοσπονδιακό χαρακτήρα, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ξεπεράσουμε τους περιορισμούς των ομόσποδων ε, κρατηδίων. Τέλος, σε σχέση με, αυτά που θίξατε, δεν ξέρω τι εννοείται όταν μιλάτε για τις ανισότητες και ως προς ένα μέσο περιφερειακό ρόλο. Εάν μιλάτε για τις ανισότητες εισόδημάτων στο εσωτερικό μιας περιφέρειας, θα ήθελα να πω ότι αυτοί οι δείκτες δεν μπορούν να υπολογιστούν. Γιατί είτε θα πρέπει να βασιστούμε σε αριθμητικά στοιχεία και κοινοτιμικές έρευνες, αλλά τα δείγματα είναι πολύ περιορισμένα, ή θα πρέπει να βασιστούμε σε δημοσιονομικές στατιστικές και εδώ υπάρχουν πολλές ε, μεροληψίες σε σχέση με τους φτωχότερους και τους πλουσιότερους. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτός ο δείκτης είναι πολύ δύσκολος να υπολογιστεί. Τι θέλετε να μετρήσετε την κοινωνική ευαλωτότητα. Εδώ υπάρχει μια σειρά άλλων δείκτων που μας επιτρέπει τις μετρήσεις αυτές, προσέχοντας το γεγονός ότι αυτοί οι δείκτες κοινωνικής ευαλωτότητας έχουν υψηλό ποσοστό μεροληψίας. Γιατί όταν μιλάμε για ανεργία θα πρέπει να δούμε, εδώ υπάρχει ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρησης. Εγώ θα ήθελα να μπορούσαμε να το κάνουμε ανεξάρτητα από τους ε, ε, δείκτες αποδοτικότητας και απόδοσης γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίος από τους μιλητές ε, μας, μας είπε το πόσο το μεγάλες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσουμε. Όμως, ο στόχος ποιος είναι. Αυτή είναι η αφετηρία μας θα πρέπει να έχουμε και κάποιους άλλους δείκτες. Εν αυτή περιπτώσει, να αναρωτηθούμε ποια είναι η ουσία αυτού του εγχειρήματο και είναι για μένα το βιωτικό επίπεδο και οπότε θα πρέπει να εξισώσουμε, θα πρέπει να υπάρχει συνοχή, θα πρέπει να υπάρχει προσέγγιση του βιωτικού επίπεδου μεταξύ των, των, των περιφερειών και θα πρέπει να, να εξαλείψουν αυτέ τι διαφορέ. Έχουμε α πούμε τι διαφορέ μεταξύ Βρυξελών, μεταξύ Βόρεια Ρενανής μεταξύ Βουλγαρίας και ο τρόπο με τον οποίο θα γίνει η μέτρηση είναι πολύπλοκο. Και έτσι θα πρέπει να δούμε πώ η ολοένα μειώμενη χρηματοδότηση απαιτεί το να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι και να ξέρουμε ρεαλιστικά τι περιμένουμε από την πολιτική της συνοχής. Ιδάλλως, δημιουργούμε προσδοκίες που δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε. Γίνεται να εξαλείψουμε, να μειώσουμε τις ανισότητες, αλλά μια που η χρηματοδότηση είναι ολένα και μικρότερη, θα πρέπει να δούμε το ότι οι περιφέρειες σύγκλησης θα εξαφανιστούν τα μέσα επόμενα χρόνια. Άρα θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να μην έχουμε στόχους μη ρεαλιστικούς. Ναι, είναι δείκτης η παινία, αλλά πώς θα τη μετρήσουμε, πώς θα την εντοπίσουμε. Νομίζω ότι αυτή η μεταβλητή είναι πάρα πολύ σημαντική. Ίσως θα μπορούσε να μετρηθεί σαν ένα ποσοστό άλλο για κάθε χώρα. Αλλά θα πρέπει να ρωτηθούμε πριν, πριν λάβουμε ένα νέο κριτήριο, να καταλήξουμε, να ρωτηθούμε με κάποιες δειγματοληπτικές μετρήσεις τι θα συμβεί. Ούτε μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όλα όσα θέλουμε. Και αυτό είναι το βασικό. Να βρούμε κάποιο κριτήριο, κάποια μεταβλητή που να είναι μετρήσιμη εύκολα, όπως τα δημογραφικά στοιχεία. Αυτό έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα σε πολλές περιοχές. Άρα το δημογραφικό είναι ίσως κάτι το χρήσιμο και επομένως έχει νόημα να έχουμε κάποιους τέτοιους δείκτες δείκτες για το εσωτερικό των κρατών μελών. Βεβαίω και υπάρχει προβληματισμό μήπω τα πράγματα χειροτερέψουν έτσι. Άκουσα προσχετικά και κατέληξα σε αυτό. Θα πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλη επιφύλαξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τους ομιλητέ για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Από πολιτική σκοπιά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η, ο, εύκολο μέθοδος είναι το ΑΕΠ. Φυσικά εδώ πολλές φορές έχουμε πει ότι δεν είναι τέλειο και πρέπει να προσπαθήσουμε να πάμε πιο πέρα. Έχουν ε, αναφερθεί διάφορες προτάσεις, διαφορετικά θέματα. Εκεί βρίσκεται το πρόβλημά μας. Υπάρχει το ΑΕΠ 1 ή το μέσο προσαρμοσμένο ή σταθμισμένο διαθέσιμο εισόδημα, αλλά βεβαίως και εδώ δεν σημαίνει ότι μπορεί κανείς να έχει το ίδιο διαθέσιμο εισόδημα από μια χώρα στην άλλη και να έχει και την ίδια αγοραστική δύναμη. Κάποια ε, χώρα, από χώρα σε χώρα αυτά διαφέρουν πολύ. Υπάρχουν οι δείκτες της ευημερίας, της φτώχειας, της υγείας, προσδοκίμου ζωής. Ε, και εδώ το προσδόκιμο ζωής δεν είναι ε, ακριβής επιστήμη γιατί ε, μερικές φορές οφείλεται στι στις συνθήκες ζωής, ε, οι συνήθειες ζωής, πολύ συχνά οι, ε, αυτοί που ευημερούν ε, είναι παχύσαρκοι, καπνίζουν κλπ. Έτσι λοιπόν εγώ θα ήθελα αυτοί οι τέσσερις ειδικοί που βρίσκονται πίσω μου να μπουν σε μια, μια αίθουσα να τους δώσουμε φαΐ και πιωτό και να καταλήξουν με έναν ορισμό του τι πρέπει να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει τόσο διαφορετικές προτάσεις. Όλες είναι λογικές σε κάποιο βαθμό, αλλά είναι σχεδόν αδύνατον να υπολογιστούν. Χρειαζόμαστε να καταλήξουμε σε μία σειρά προτάσεων. ΑΕΠ συν 1, συν 2 ή κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ρίκα, σε παρακαλώ στο πιο σύντομα. Ευχαριστώ πράγματι. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Καταρχήν, νομίζω ότι το ΑΕΠ χρειάζεται κάτι άλλο, έναν συνοδευτικό δίκτυο δηλαδή. Δεν σημαίνει όμως ότι το ΑΕΠ είναι και το πιο σημαντικό κριτήριο. Ακούσαμε πολλά επιχειρήματα υπέρ της ύπαρξης άλλων κριτηρίων. Εάν λάβουμε υπόψη το ΑΕΠ καθεαυτό δεν αντικατοπτρίζει τα ουσιώδη πρόβλημα που υπάρχουν στους ε, μεμονωμένους ε, τομείς. Όπως ακούσαμε και στις ε, παρουσιάσεις, πολλές φορές ισχύει κάτι τέτοιο. Όταν μιλάμε λοιπόν για ύπαρξη δικτών, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι θα πρέπει να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ των διαφόρων τομέων και πώς μπορεί να υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο και αποδοτικό για τους ανθρώπους. όταν είπατε, όπως είπατε, αρχίζουμε με αρνητικές δίκ, δείκτε, δείκτες και αυτό δεν μας υποστηρίζει, δεν υποστηρίζει την κατάσταση. Ίσως θα πρέπει να αρχίσουμε με κάτι πιο θετικό, δηλαδή όταν ξεπερνάμε ένα κατόφλι, τότε υπάρχει μια θετική ροπή. Επίσης θα πρέπει να μετράμε τα βιώσιμα αποτελέσματα. Θα ήθελα να πω και κάτι άλλο ως προς το δημογραφικό ζήτημα και τη γύρανση. Όταν μιλάμε για νέους δείκτες Νομίζω ότι ως προς τη μέτρηση αυτή είναι μια θετική λύση γιατί η γύρανση έχει αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα και θα έπρεπε να μπορέσουμε κάτι να κάνουμε, αυτό, ε, κάτι να κάνουμε γι' αυτό αρχικά ως προς την περιφερειακή πολιτική. Επίσης, ως προς τη, τη ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχει μεγάλη σημασία να δούμε πώς ορίζουμε τις πόλεις στα αστικά κέντρα, γιατί υπάρχουν μεγάλες διαφορές στη Φιλανδία. Έχουμε πολλές πόλεις κάτω των 100.000 κατοίκων, αλλά διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν καλύτερους δείκτες που να αντικατοπτρίζουν τα προβλήματα καθώς και τους αντικτύπους. Ε, τέλος, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να ε, προσθέσετε κάτι από πλευράς ε, ε, Κομισιόν. Σύντομα παρακαλώ. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μία σοβαρή πτυχή. Θα πρέπει να συγκρίνουμε μεταξύ ε, βημάτων για τη σύνταξη μιας πολιτικής συνοχής. Θα πρέπει να επιλέξουμε τις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες, να δούμε πώς έχει η χρηματοδοτική κατανομή και τέλος να ορίσουμε τα ίδια τα προγράμματα καθεαυτά. Ως προς την επιλεξιμότητα νομίζω ότι χρειαζόμαστε δείκτες ε, που εμπεριέχουν ορισμένα στοιχεία, στοιχεία χρονικής σταθερότητας. Θα πρέπει να υπάρχει συνένεση ως προς το περιεχόμενο των δικτών και ε, επίσης ε, θα πρέπει οι πόροι να πηγαίνουν προς τις μειονεκτούσες και φτωχότερες περιοχές, γιατί αυτό είναι ο βασικός στόχος της πολιτικής συνοχής. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχει εναρμόνιση σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτό μειώνει τις επιλογές μας ως προς τους δείκτες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως προς την κατανομή. Μην ξεχνάτε ότι ενσωματώνουμε και άλλους δείκτες σε σχέση με την κατάρτιση, περιφέρεια και οι εμπλεκόμενοι φορείς και τα θεσμικά όργανα, οι περιφέρειες, οι τοπικές αρχές ορίζουν τα επιχειρησιακά προγράμματα. Γιατί εδώ έχουμε πληθώρα δικτών που λαμβάνονται υπόψη και άρα κινούμεθα πέραν του ΑΕΠ. Ευχαριστώ τώρα οι πάνελιστοι, οι εμπειρογνώμονες. Κάτι πρέπει να μας πούν. Ναι. να προσθέσω κάτι σε αυτά τα τρία βήματα είναι το να ενημερώνει κανείς το κοινοβούλιο, να υπάρχει feedback και έτσι να προετοιμάζει ο τάδος για τις επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές. Επίσης και την ισότητα των φίλων να λαμβάνει υπόψη για τους δείκτες. Ε, δεν βλέπετε εδώ πέρα, γιατί το λέω αυτό, γιατί εδώ είμαστε τέσσερις άντρες. Επαναλαμβάνω ότι οι δημογραφικοί δείκτες είναι κατανοητοί και μετρήσιμοι. Άρα θα πρέπει να περιληφθούν και αυτοί. Εσείς καθηγητά, Φάντερμαν, δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτα-πρώτα να καθισχάσω τον κύριο Κέλλη ότι όσον αφορά το εισόδημα λαμβάνει υπόψη αγροτική δύναμη αλλά όχι περιφερειακά, εθνικά. Δεν είναι το ίδιο. Είπε κάποια κυρία ότι ο στόχος θα πρέπει να είναι οι διαφορές οι μικρότερες μεταξύ των περιφερειών. Ξαρτάται τι επιδιώκει κανείς. Θα μπορούσε κανείς να έχει ως στόχο σε μια χώρα να έχει έναν άδειο χώρο όπως ένα πάρκο και κάπου αλλού που να έχει συγκεντρωμένη οικονομική δραστηριότητα. Είναι θέμα πολιτικής επιλογής. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή η μικρότερη διαφορά μπορεί να είναι ένας δείκτης όπως το διαθέσιμο εισόδημα. Γιατί εκείνοι που μένουν σε μια περιφέρεια όπου έχουμε στόχο του να κάνουν αυτή την περιοχή φυσικό πάρκο, ότι θα πρέπει να έχουν ένα βιωτικό επίπεδο συγκρίσιμο με την υπόλοιπη χώρα. Όμως, τι θα πει συνοχή, ότι θα πρέπει να υπάρχει ομοιομορφία παντού, είναι αυτό το ένα ερώτημα στο οποίο η πολιτική θα πρέπει να απαντήσει ή να απαντήσουν οι πολιτικοί. Η γύρανση του πληθυσμού δείκτης και εν προκειμένου ο κάθε δείκτης συνδέεται με το τι επιδιώκει κανείς. Μπορούσε κανείς να πει ότι το είναι καλό και είναι κακό. Εδώ θεωρούμε ότι οι γεννήσεις έχουν πέσει και από την άλλη μεριά άλλωστε μπορείς να θεωρήσει ότι είναι καλό κακό μόνο ότι έχουν μειωθεί οι γεννήσεις και καλό διότι τώρα έχουμε περισσότερους ηλικιωμένους. Και άρα κανείς ζει περισσότερο. Επομένως, η επιλογή ανήκει στους πολιτικούς. Η γύρανση επίσης δημιουργεί και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ευτυχώς σήμερα δεν καλούμεθα να αποφασίσουμε για τους δίκτυες αλλά νομίζω ότι αυτή η συζήτηση και ιδίως αυτά που μας είπατε, μελέτες, έρευνες, εμπειρία σας, όλα αυτά νομίζω μας άνοιξαν καινούριου δρόμους για να προβληματιστούμε και στις διαπραγματεύσεις μας για το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ευχαριστώ. Ευχαρίστως. Διαβιβάστε μας ε, τα έγγραφα με τις ε, σκέψεις σας. Ήδη έχουμε κάποιο υλικό. Έχω να πει για την Κομισιόν ότι βεβαίως και από εσάς θα χρειαστεί να έχουμε στοιχεία και να συζητήσουμε ό,τι από το ρυθμιστικό κανονιστικό πλαίσιο έχει να κάνει με τους δείκτες. Συνάδελφοι, εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας. Δεν έχουμε διάφορα εκτός αν εσείς έχετε κάτι να προτείνετε για τα διάφορα. 25 πρώτο θα συνδεθούμε. Θέλω να σας ευχηθώ και πάλι. Καλή ξεκούραση για τις επόμενες δύο εβδομάδες που δεν θα βρισκόμαστε σε αυτό το κτίριο. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς και εσείς τις καλύτερες ευχές. Καλή χρονιά. Uh, thank you very much. Um, and the meeting is adjourned. Πέρα